Ναι, πες Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να επαναλάβουμε τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα εκ μέρους σας να χαιρετήσω την Επίτροπο που είναι αρμόδια για τα θέματα υγείας, την κυρία Ανδρούλα Βασιλείου. Είναι φυσικά ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει και στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα του της νέας γρήπης. Βρισκόμαστε στην απαρχή της νέας νομοθετικής ε, περίοδου. Έχουμε πολλά μέλη τα οποία είναι ενθουσιώδη και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα και για τα θέματα του περιβάλλοντος και για τα θέματα της υγείας που είναι από τις πρώτες προτεραιότητές τους και η στενόπιόν μας σήμερα για να μας παρουσιάσετε την κατάσταση της αντιμετώπισης του ιού H1N1 ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα την ε, κοινή γνώμη. Η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ήδη ότι θα έχει ένα πρόγραμμα για τα θέματα αυτά που θα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα γνωρίσουμε τις λεπτομέρειές του. Έχουμε στη διάθεσή μας 1,5 ε, μια μισή ώρα και θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να είναι περιορισμένοι στη χρήση του λόγου. Η κυρία Επίτροπος έχει πρώτα το λόγο. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι ιδιαίτερος που για πρώτη φορά μετά τις ευρωεκλογέ έρχομαι στην Επιτροπή σας. Πρέπει να πω ότι είχα πολύ καλές σχέσεις με την Επιτροπή σας στην προηγούμενη θητεία και πιστεύω ότι η καλή σχέση θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Όπως είπε και ο πρόεδρός σας, μου ζητήθηκε να έρθω και να σας κάνω μία παρουσίαση για το τι κάναμε τους τελευταίους μήνες σε σχέση με την πανδημία H1N1. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω πως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και μετά να σας μιλήσω για τις προσπάθειές μας που συνεχίζονται για τη διαχείριση και περαιτέρω προετοιμασία. Σήμερα όλες οι χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΖΕΣ έχουν αναφέρει επιβεβαιωμένες ε, περιπτώσεις, ε, κρούσματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερα από 55.000 κρούσματα στην Ευρώπη, όμως πολλές χώρες έχουν σταματήσει πλέον να μετράνε, άρα το νούμερο δεν είναι αξιόπιστο, νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο και παγκοσμίως έχουμε περίπου 350.000 κρούσματα. Όπως είπα όμως, αρκετές χώρες έχουν σταματήσει να αναφέρουν τα νούμερα, οπότε μάλλον τα νούμερα είναι μεγαλύτερα. Ο ρυθμός μόλυνσης είναι μεγαλύτερος στην ηλικία μοάδα 5 έως 24 ετών, ενώ στο νοσοκομείο καταλήγουν περισσότερα άτομα στην ηλικιακή ομάδα μέχρι 4 ετών. Παρ' όλα αυτά, οι περισσότερες ε, περιπτώσεις είναι με ήπια συμπτώματα, ωστόσο έχουμε περίπου 170 θανάτους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Αν και η πλειονότητα των θυμάτων είναι άτομα που ήδη είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών, οι θάνατοι παγκοσμίω είναι περίπου οι ίδιοι με αυτούς της εποχικής γρήπης που όσο γνωρίζουμε κάθε χρόνο σκοτώνει 250.000 με 500.000 άτομα. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η πανδημία αλλά και η εποχική γρήπη είναι αυλαβής. Με βάση την τρέχουσα ανάλυση για τη συμπεριφορά της πανδημίας στο νότιο ημισφαίριο, η CDC e εκτιμά ότι στην χειρότερη περίπτωση μέχρι 30% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αμολυνθεί με τον ιό κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος ότι με την πάροδο του χρόνου ο ιός ε, της γρήπης θα μεταλλαχθεί και θα γίνει περισσότερο παθογόνος. Σε μια τέτοια περίπτωση τα αποτελέσματα της μόλυνσης μπορεί να είναι πλέον πιο σοβαρά. Αυτό θα σήμαινε μεγάλη, τεράστια πρόκληση από πλευράς διαχείρισης δημόσιας υγείας και θα σήμαινε επίσης και μεγάλο βάρος για τις υγειονομικές υπηρεσίες και γενικά για την οικονομία. Πρέπει να θυμούμαστε ότι οι πανδημίες γρήπες είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Όμως πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι έτσι ώστε να μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειες της πανδημίας. Βεβαίως, οι τεχνικές δυνατότητες οι οικονομικές δυνατότητες και η ετοιμότητα δεν είναι ίδιες σε όλα τα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη είναι πιο καλά προετοιμασμένα για τη διαχείριση της κατάστασης. Γι' αυτό χρειάζεται μία συντονισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στην κρίση. Τα τελευταία χρόνια τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν σχέδια εθνικής ετοιμότητας με έμφαση στο συντονισμό της πρόληψης και των μέτρων ελέγχου και την αύξηση των δυνατοτήτων αντιμετώπισης μια πανδημίας γρήπης. Πριν παλαιότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε θεωρήσει ότι είναι προτεραιότητα η ετοιμότητα για μια γρήπη το Νοέμβριο του 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σχετική ανακοίνωση για την ετοιμότητα για πανδημίες γρήπης και αυτή περιέχει διάφορα εργαλεία και μηχανισμούς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη. Από τότε που ξεκίνησε τον Απρίλιο η πανδημία, τα κράτη-μέλη έχουν συντονίσει τις προσπάθειές τους με βάση τον σχεδιασμό ετοιμότητας που είχαν ήδη κάνει. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ηγείται των προσπαθειών συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις Μεταδοτικές Ασθένειες και τα συμπεράσματα του έκτακτου Συμβούλιου Υγείας της 30 Απριλίου. Προκειμένου να διαχειριστούμε το συντονισμό, εγώ ενεργοποίησα το HEOF της Επιτροπής, το οποίο θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα ηγείται κοινών συναντήσεων μεταξύ των αρχών δημόσιας υγείας των κρατών μελών. Η Κομισιόν στηρίζεται στο έργο της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας στην οποία συμμετέχουν αξιωματούχοι υψηλού επίπεδου από τις εθνικές κυβερνήσεις. Είναι ένα άτυπο όργανο συνεργασίας και συντονισμού που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή πληροφοριών για απειλές της υγείας. Από το ξεκίνημα της πανδημίας είχαμε μέχρι 30 τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους από τα κράτη-μέλη καθώς και άλλες συναντήσεις με εκπροσώπους τρίτων χωρών και του ΠΟΗ. Στέλνουμε τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων στους διάφορους ενδιαφερόμενους ενώ επίσης συνοπτικά πρακτικά μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΓΔ ΣΑΝΚΟ. Αυτή τη στιγμή έχουμε συναντήσεις ε, μία φορά την εβδομάδα και επικεντρωνόμαστε κυρίως σε θέματα διαχείρισης κινδύνου. Χάρη στην προσπάθειά μας για το συντονισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει σειρά μέτρων για την καλή διαχείριση της πανδημίας, όπως κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση των κρουσμάτων και τις θεραπείες και για την συμβουλές για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν τα ιατρικά. Συμβουλές στο κοινό για την, τα προσωπικά μέτρα προστασίας, δηλώσεις όσον αφορά το κλείσιμο σχολείων, ε, της ομάδας προτεραιότητας και ταξιδιωτικές οδηγίες και τέλος έναν κοινό ορισμό του TST κρούσμα για την καλύτερη διάγνωση. Εδώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμφώνησε στις αρχές του έτους να επιταχύνει τις διαδικασίες που μας επιτρέπουν να εγκρίνουμε ορισμούς κρουσμάτων για τον H1N1. Αν επαναληφθεί αυτή η ανάγκη εντός του φθινοπόρου. Ελπίζω ότι θα έχω ανάλογη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αντιμετωπίσουμε άμεσα την κατάσταση. Προκειμένου να ενισχύσουμε το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων τομέων και μεταξύ των κρατών μελών, στις 15 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μία ανακοίνωση που συγκεντρώνει όλα τα βασικά θέματα και όλες τις βασικές απαντήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε μία μόνη έκθεση. Η ανακοίνωση έχει τρεις στόχους. Πρώτον, αναφέρει τα βασικά επιτεύγματα της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την αρχή της επιδημίας. Όπως το ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν πρόσβαση στις τελευταίες επιστημονικές συμβουλές και τεχνικές συμβουλές μέσω ευρωπαϊκών οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Επίσης, υπάρχει συμφωνία όσον αφορά κοινέ προσεγγίσεις για το κλείσιμο σχολείων, τις ταξιδιωτικές οδηγίες, τους ταξιδιώτες με συμπτώματα και της ομάδας προτεραιότητες για τα εμβόλια. Ο δεύτερος στόχος αφορά πιο ευρεία θέματα που έχουν να κάνουν με την διατομεακή συνεργασία και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Και ο τρίτος στίχος αφορά τα πιο συγκεκριμένα προβλήματα, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη εμβολίων και αντιακών, η προμήθεια εμβολίων και οι στρατηγικές εμβολίων, η παροχή στήριξης για τρίτες χώρες και η αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού. Αυτά τα συγκεκριμένα θέματα αναφέρονται με λεπτομέρειες στα πέντε έγγραφα εργασίας που συνοδεύουν την ανακοίνωση. Αυτό το πακέτο λοιπόν θα αποτελέσει τη βάση των συζητήσεων της έκτακτης συνεδρίασης των Υπουργών Υγείας στις 12 Οκτωβρίου. Προκειμένου να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στην πανδημία, συνεργαζόμαστε και με βασικούς εταίρους παγκοσμίω. Στις 11 Σεπτεμβρίου ηγήθηκα της ε, Υπουργικής Συνάντησης ε, για την ε, Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ασφάλειας Υγείας που, όπου συμμετείχαν οι χώρες του G7 και το Μεξικό. Ασχοληθήκαμε κυρίως με τον εμβολιασμό και την παροχή στήριξη σε τρίτες χώρες. Αυτή η ομάδα παρήχε πολύ χρήσιμη συμβολή για την διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό. Περνάω τώρα στο πολύ σημαντικό θέμα των εμβολίων. Την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΜΕΑ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων γνωρίζω ότι θα συναντηθείτε σήμερα με τον διοικητή της ΕΜΕΑ. Η ΕΜΕΑ λοιπόν δημοσίευσε θετικές γνωμοδοτήσεις που συνιστούν τα δύο εμβόλια που υπάρχουν και ζήτησε να αδειοτηθούν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Λόγκρεν θα σας μιλήσει αργότερα για αυτά. Και εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης των αδειοδοτήσεων αυτών των εμβολίων. Επίσης, η Κομισιόν έχει κάνει συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη στρατηγική εμβολιασμού και τον εντοπισμό των ομάδων προτεραιότητας. Αυτές οι συστάσεις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Ασφάλειας Υγείας με στόχο να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των στρατηγικών για τον εμβολιασμό τους. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητά αξιότιμα μέλη, οι συνέπειες από την πανδημία μέχρι στιγμής είναι σχετικά περιορισμένες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να λάβουμε τις μέγιστες δυνατές προλήψεις για την αντιμετώπιση αυτού του νέου ιού γρήπης, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι αυτή η ιή. Στις 11 Σεπτεμβρίου που συναντηθήκαμε με τους διεθνείς εταίρους, θυμάμαι πολύ καλά τι είπε ένας εμπειρογνώμονας του ΠΟΗ. Κανείς, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πώς θα εξελιχθεί αυτός ο ιός. Μπορεί να παραμείνει ελάσσονος σημασίας όπως τώρα, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ πιο σοβαρός και όλοι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το ενδεχόμενο. Σίγουρα είμαστε καλά προετοιμασμένοι, αλλά πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή καθώς έρχεται ο χειμώνας για να είμαστε σίγουροι ότι είναι προστατευμένοι οι πολίτες μας και ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τα κατάλληλα μέτρα. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα μπορώ να βασιστώ στην πολύτιμη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικά της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, κυρία Βασιλείου, για την παρουσίασή σας και για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη για να είναι πράγματι προπαρασκευασμένη ενώπιον της ε, γρήπης αυτής η οποία έχει μεγάλη, ε, μεγάλη, έχει λάβει μεγάλη έκταση και δεν πρέπει να βρεθεί εκτός έλεγχου βρισκόμαστε στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητος και εγώ ο ίδιος ε, εμβολιάστηκα εναντίον της ε, γρήπης και ξέρετε το Κοινοβούλιο δίνει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν. Φυσικά αυτό είναι ένα θέμα προσωπικής απόφασης. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχουν τα εμβόλια για, τις, ε, για την αντιμετώπιση της γρήπης και νομίζω ότι όλα αυτά τα έχουν εξετάσει και τα έχουν εγκρίνει οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη. Τώρα, οι ομιλητέ ξεκινούμε με τον κύριο Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο για την τόσο χρήσιμη αυτή παρουσίασή της και τη δέσμευσή της για το θέμα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Κομισιόν να παίξει το συντονιστικό ρόλο και να είναι αρρωγός των κρατών μελών στην αντιμετώπιση της γρήπης γιατί πρόκειται για μια πανδημία και κανεί δεν θα κατανοούσε το να ακολουθήσει η Κομισιόν μια στάση η οποία δεν ήταν συνεκτική με αυτή των κρατών μελών και θα είχαμε διαφορετικές πολιτικές σε κάθε κράτος μέλος. Εγώ επίσης χαίρομαι για το γεγονός ότι δόθηκε αυτή η σύσταση σε σχέση με το κλείσιμο των σχολείων μετά από τη συζήτηση που έχει γίνει στα κράτη-μέλη. διακόπτε το ομιλητής. Η Βραζιλία κατά την άποψή μου είναι κατά τις πληροφορίε που έχω μάλλον είναι η χώρα που είχαν γίνει τα περισσότερα θανατηφόρα κρούσματα και κλείσαν τα σχολεία πριν από τρεις εβδομάδε. γιατί τα παιδιά ουσιαστικά προσελκύονται από τα καταστήματα που είναι έξω από τα σχολεία και δεν πηγαίνουν να εμβολιαστούν και να έχουν την κατάλληλη αντιμετώπιση να, να... να προλάβουν την ε, ασθένεια αυτή. Τώρα για τα αντιϊκά φάρμακα, από ό,τι γνωρίζω, η έγκριση αφορά όλες τις ομάδες του πληθυσμού ε, και τις ομάδες πληθυσμού που είναι ομάδες κινδύνου επίσης και ε, αυτές οι οποίες είναι τις ομάδες των παιδιών. Η εκπρόσωπος του Οργανισμού για την Πρόληψη των Ασθενειών ανέφερε ότι αυτό αφορά και τους ενήλικες. Ε, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει ακόμα σαφήνεια για το θέμα αυτό γιατί απλώς υπήρξε η έγκριση ενός δείγματος και όχι συνολική έγκριση. Πάντως υπάρχει η σύσταση να εμβολιάζονται πρώτα τα παιδιά και θα ήθελα λοιπόν να έχω κάποια διευκρίνηση από εσά για το αν θα μπορούσε να γίνει το ταχύτερο δυνατόν ο εμβολιασμό των παιδιών και των ομάδων κινδύνου. Δεύτερον, για τα φάρμακα αυτά έχω τις πληροφορίες ότι Υπάρχει αρκετή ποσότητα ταμιφλού αυτή τη στιγμή για τον εμφυβολιασμό αυτό και επειδή και η κυρία ε, Γκρόστατ είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για το θέμα αυτό, νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί πλήρως. Τώρα η τελευταία μου παρατήρηση δεν μου είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Ε, δεν είναι σαφές τώρα, μέσα στη διαδικασία αυτή, της έγκρισης των φαρμάκων αυτών, αν αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Ο πρόεδρος ε, και ποιος θα είναι ο επίτροπος ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Ο κύριος ε, ε, Μπαρόσο θα πρέπει να αποφασίσει ποιος θα αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αλλά, κυρία Βασιλείου, αν σας ζητήσει ο κύριος Μπαρόσο αν τα θέματα αυτά θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστούν από ένα άλλο επίτροπο εκτός από τον Επίτροπο Υγείας, θα έχετε μια θετική ή μια αρνητική άποψη. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Είναι παρόν ο κύριο Λούντγκεν, ο εκτελεστικός διοικητή της ΕΜΕΑ, του Φορέα για τα Φάρμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Και νομίζω τα ειδικά θέματα θα ήταν καλύτερα οι συνάδελφοι να τα απευθύνουν στον κύριο Λούντγκεν για να μην έχουμε επικάλυψη και να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα τι λεπτομέρειε που αφορούν τους ειδικού να τις συζητήσουμε αργότερα το απόγευμα. Κυρία Ροτ Μπέρεντ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα που θα συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Λέγκριν σήμερα, όπω είπατε και εσεί, εκεί όπου θα συζητήσουμε τη διαδικασία έγκριση για τα εμβόλια. Και δεν θα ασχοληθώ επίση και με το ζήτημα ε, του κατά πόσο τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι καθαρά θέμα υποφόρα την υγεία ή και ε, ε, άλλα θέματα εμπορικά. Κύριε πρέπει να σα πω ότι πάντα σα ακούω, εντυπωσιάζομαι. Τι γίνεται όμω, μετά πάω σπίτι μου ή πάω σε μια άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και χάνω αυτό το πρώτο μου συνέστημα. Μιλήσατε για όλες αυτές τις συνεδριάσεις που κάνατε, 30 όντιο συνδιασκέψεις. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι συμμετέχοντες είναι ε, οι πλέον οι, οι δήμονες. Αλλά κοιτάξτε να σας πω το εξής. Εξακολουθώ να βλέπω να λείπουν ορισμένα πράγματα τα οποία τα είπα και όταν, είπε, και όταν ήταν η κυρία Τζέικοψον. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το θέμα τη πληροφόρηση. Εξακολουθώ να βλέπω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη ήταν λίγε οι πληροφορίε που δόθηκαν, δεν ήταν συνεπεί δεν ήταν ε, οι ίδιε πληροφορίε και, στην ίδια, και σε ίδιο σημείο. Δηλαδή, δεν δόθηκαν σε κάθε σχολείο, σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε ε, πόρτα γραφείου, σε κάθε διοικητική υπηρεσία και εκεί δεν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες. Να ε, ε σφίγγουν το χέρι του συνανθρώπου τους, ε, να ε, αποφεύγουν το μετρό. Τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Εδώ μιλάμε για απλούστατες πληροφορίες. Αν μέσα από όλες αυτές τις συνδυάσεις δεν μπορούμε να έχουμε αυτό αποτέλεσμα, ε, τότε τι να πω. Και τώρα, έχουμε το δεύτερο θέμα, προφύλαξη. Με εξέπληξε ιδιαίτερα όταν αρχίσαμε τα σχολεία πάλι το Σεπτέμβριο, τέλος Αυγούστου ή Σεπτέμβριο ανάλογα με τη χώρα, και με εξέπληξε το γεγονός ότι ε, δεν ήταν διαθέσιμο, διαθέσιμο παντού υλικό για απολύμανση των χεριών. Δεν ήξεραν όλοι τι πρέπει να κάνουν. Ε, για παράδειγμα, ε, ε, τι να κάνουμε τον καφέ. Το γράφουν ορισμένε εφημερίδες, αλλά δεν είναι παντού γνωστό. Για παράδειγμα ότι άμα δεν έχει άλλη δυνατότητα να απολυμάνει τουλάχιστον τα χέρια σου, έστω και με ε, η, Τέλο πάντων, μια σειρά από προφυλάξει που θα έπρεπε να δίδονται πληροφορία. Ετοιμότητα και συμβουλή, τα άλλα δύο θέματα. Ετοιμότητα. Το ξέρουμε, εντάξει. Και σήμερα είχαμε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό ε, για την ετοιμότητα ε, και αυτόν τον ενθουσιασμό που έχουν τα καινούργια μέλη. Ε, ψηφίσαμε σήμερα στον προπολογισμό για στήριξη των κρατών μελών για να αγοράσουν τα αντίοικα και τα εμβόλια. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ότι δεν έχει καμία σχέση με τον προπολογισμό, τέλο πάντων τα ψηφίσαμε. Άλλο θα γίνει στην Ολομέλεια. Α το ξαναπούμε. Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και ρωτώ, είναι έτοιμα. Και αν δεν είναι έτοιμα, γιατί. Αρχι... Μπορούμε να αρχίσουμε να κατονομάζουμε κυρία Βασιλείου. Σα παρακαλούμε. Έχουμε μια κάπω μια χοντρική ιδέα για το τι γίνεται στη χώρα μα. Μήπω θα μπορούσαμε, σα παρακαλούμε, να σχηματίσουμε μια εικόνα ε, τι γίνεται σε, σε τα κράτη-μέλη, ε, νοσοκομιακές κλίνες, ε, αντιϊκά εμβόλια, τι ακριβώς γίνεται στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι η ετοιμότητα. Τελειώνω, τελειώνω βέβαια. Και μετά στο θέμα της Συμβουλής. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε στους πολίτες τι να κάνουν δεν ξέρουν τι να κάνουν, να εμβολιαστούν ή να μην εμβολιαστούν. Ε, αυτό πρέπει να του το δώσουμε εμεί ω συμβουλή και πρέπει να δοθεί σε κάθε κράτο μέλο. Δεν ξέρουν τι να κάνουν οι πολίτε. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε τον κύριο Λάγκεν ε, το είδο του υλικού που έχουμε, αλλά αυτό δεν, είναι, δεν αρκεί. Δεν είναι ε, δουλειά του οργανισμού για τα φάρμακα να ασχοληθεί με αυτό και μόνο. Ε, σας παρακαλώ μπορείτε να μα βοηθήσετε στο σημείο αυτό. Θέλετε να απαντήσετε, ναι. Κοιτάξτε, συμφωνώ μαζί σας. Ευθύνη μας είναι να φροντίσουμε έτσι ώστε όλα τα κράτη-μέλη θα έχουν τις ίδιες πληροφορίες, θα έχουν πάρει από εμά τις ίδιες κατευθυντήρες γραμμές, την ίδια συμβουλή και να, συν, και να συμφωνήσουμε σε ένα ενιαίο τρόπο ε, κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών στου πολίτε. Αλλά το ξέρετε. Αν προσπαθήσω να κάνω κάτι περισσότερο από αυτά και να αρχίσω να ρωτάω ερωτήσει στους υπουργού, τι κάνατε για το Α, για το Β, ε, όλοι θα με κατηγορήσουν για επέμβαση στις δικές του αρμοδιότητες. Το ξέρετε. Η θέση μου είναι πολύ λεπτή λοιπόν. Προσπαθούμε και δίνουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Συμφωνούμε σε ορισμένα έγγραφα πώς να έρχομαι σε επικοινωνία με τους πολίτες, με το κοινό, τι θα γίνει με το κλείσιμο των σχολείων, με τις συμβουλές προς ταξιδιώτες. Τα έχουμε συμφωνήσει όλα αυτά. Αλλά σε τελευταία ανάλυση οι Υπουργοί υγεία είναι αρμόδιοι για να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Οι Υπουργοί υγεία, λοιπόν ε, έχουν διακριτική ευκαιρία να τα ακολουθήσουν ή να μην τα ακολουθήσουν. Βεβαίω, αύξηση τη τοποίηση του, του κοινού. Γιατί τώρα, όταν εγώ ταξιδεύω στα κράτη-μέλη, βλέπω το εξή. Έρχονται ορισμένοι και με ρωτούν. Είναι τελικά τόσο σοβαρή η κατάσταση. Γιατί δεν το συζητά κανεί το θέμα. Μήπω ε, δεν χρειάζεται να προσέχουμε αυτά τα ζητήματα. Ε, Ακριβώ γι' αυτό. Α πιέζω του υπουργού υγεία να διατηρήσουμε την επαγρύπνησή μα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. σω τελευταία ανάλυση μα κατηγορήσουν ότι κάναμε περισσότερα από ό,τι χρειαζόταν. Ε, τι να σα πω, δεν μπορούμε να κερδίσουμε ποτέ. Καλύτερα να μα κατηγορήσουν ότι κάνουμε πολλά παρά να μα κατηγορήσουν ότι απέναντι στι σοβαρέ εξελίξει δεν ήμασταν έτοιμοι. Είναι αλήθεια. Ότι είχαμε πάνω από 30 βίντεο συνδιασκέψεις με εκπροσώπους των κρατομελών. Συμφωνήσαμε σε πολλά ζητήματα. Αλλά τι να σας πω, ε, είναι δική του αρμοδιότητα των κρατών μελών να τα εφαρμόσουν όλα αυτά. Κυρία Corinne Η Κορίν Λεπάζ. Κύριε Επίτροπε, εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά όλα αυτά τα ερωτήματα, τα δύσκολα τα οποία τίθενται λόγω της ε, αρχής της επικουρικότητας. Αλλά όπως σας έλεγε και ο κύριος Λίζε προηγουμένως, εμείς πριν από μερικές εβδομάδες ακούσαμε την κυρία Γέρκαπ, η οποία μας είπε σαφώς ότι τα εμβόλια αυτά όταν θα είναι διαθέσιμα και εφόσον υπάρχει η έγκρισή τους αφορούν τα ενήλικα άτομα που είναι σε καλή υγεία. Ενώ τα εμβόλια που αφορούν τα άτομα σε ομάδες κινδύνου και τα παιδιά, αυτά ήταν μια διαφορετική υπόθεση. Γιατί η μελέτη για τα δυνητικά αποτελέσματα αυτών των εμβολίων θα ξεκινήσει μονάχα τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά από την θέση σε εμπορία των πρώτων αυτών εμβολίων. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτή είναι η θέση που έχει υιοθετήσει η Κομισιόν για το θέμα αυτό, γιατί κάπως με, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά. Το γεγονός δηλαδή ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη λέμε ξεκινάμε με τα παιδιά και τα άτομα που είναι ομάδες, στις ομάδες κινδύνου, ενώ, ενώ η στάση της κυρίας Γιακάμπη ήταν περίπου η αντίθετη από αυτήν τη στάση. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα το οποίο που ετέθηκε από την κυρία Ριβαζή προηγουμένως είναι το θέμα της σύνθεσης αυτών των ε, φαρμάκων και των στοιχείων που περιέχονται σε, αυτήν, σε αυτά τα φάρμακα. Είναι ίσως ένα τεχνικό θέμα το οποίο πρέπει να θέσουμε στον εκπρόσωπο της ΕΜΕΑ, της ε, ε, υπηρεσίας για τα φάρμακα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι. Ποια είναι τα συνέκδοχα τα οποία περιέχουν τα φάρμακα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι τα αρνητικά αποτελέσματα αυτών των φαρμάκων δεν θα είναι σημαντικότερα από το θετικό αποτέλεσμά τους. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί από τους συμπολίτε μας και γι' αυτό σας το θέτω. Θα το θέσουμε το ερώτημα αυτό στον κύριο Λούντρια. Λοιπόν, θα μαζέψουμε ορισμένε ομιλίε, ορισμένε παρεμβάσει, ερωτήσει και θα απαντήσετε στη συνέχεια η Γκροστέτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> κύριε Επίτροπε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε πάντα στην Επιτροπή αυτή. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία είναι θέματα αρμοδιότητας του Διευθυντή του, της Υπηρεσίας Φαρμάκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς θέλω να σταθώ στην ανάγκη να υπάρχει σωστή επικοινωνία, γιατί βλέπω ότι ακόμα και στα κρατημέλη όπου υπάρχει καλή επικοινωνία εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, εξακολουθεί να υπάρχει πλήρης σύγχυση. Σύγχυση μεταξύ εποχικής γρήπης και της ε, γρήπης του ιού H1N1. Γιατί λέει πολλοί κόσμοι η εποχική γρήπη εντάξει δεν είναι κάτι το τρομερό, τόσοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο, αν τελικά η H1N1 είναι παρόμοια με την εποχική γρήπη γιατί κάνουμε τόση φασαρία. Αυτό όμως μου φαίνεται ότι είναι επικίνδυνη στάση εν ώψη των πληροφοριών που έχουμε, ότι δεν ξέρουμε καθόλου πώς μπορεί να μεταλλαχθεί ενδεχομένως αυτός ο ιός από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να, κάνουμε, να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. Πώς λοιπόν κύρια Επίτροπε προβλέπετε να αντιμετωπίσετε αυτές τις κριτικές, παραδείγματος χάρη σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτά τα φάρμακα. Υπήρξαν πολλοί ιατροί οι οποίοι λένε ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Λένε άλλοι ότι υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού που πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα. Πώς θέλετε λοιπόν ο πληθυσμός να ξέρει τι γίνεται όταν λένε οι ίδιοι παθολόγοι ότι δεν είναι χρήσιμο το φάρμακο και δεν πρόκειται το εμβόλιο και δεν πρόκειται να εμβολιαστούν. Όλα αυτά λοιπόν είναι για μένα πολύ επικίνδυνα, επικίνδυνες πληροφορίες για την κοινή γνώμη, γιατί αν το χειμώνα <clears throat> προκύψει κάποια σοβαρή πανδημία με μια τροποποίηση και μετάλλαξη του ιού και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό θανάτων, τότε ο πληθυσμός θα περάσει σε κατάσταση τρέλας και παραλογισμού και θα είναι πολύ αργά πια για να τον εμβολιάσουμε. Βέζιχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω αρκετές ερωτήσεις. Καταρχάς όσον αφορά τις εγκρίσεις. Με εκπλήσει ότι δεν ξέρω, εγώ είμαι εκλεγήθησα, αλλά βλέπω ότι Υπάρχει μια περίεργη διαδικασία έγκρισης. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα είναι η Επίτροπος που θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση. Δεύτερον, βλέπω ότι δεν υπάρχουν κλινικά δεδομένα για τις έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. Όλα τα δεδομένα που έχουμε είναι προβολές με βάση το make-up. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε αυτό το εμβόλιο και χρησιμοποίησαμε δεδομένα από άλλο στέλεχος του h n 1 Επίσης, δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία για παιδιά μέχρι τριών ετών, πολύ λίγα για την ηλικία ομάδα 3-10 ετών και καθόλου δεδομένα για τις έγκυους γυναίκες. Όμως, για ποιους θεωρούμε ως μεγαλύτερες προτεραιότητες τα παιδιά με προβλήματα άσθματος και τις έγκυους γυναίκες. Δεύτερον, θέμα ευθύνης. Χτες ήρθα σε επαφή με το εργαστήριο της Νοβάρτης, στους οποίους πρόκειται να δώσετε έγκριση. Και στο ερώτημά μου, ποιος θα είναι υπεύθυνο αν προκύψουν παρενέργειες μετά τον εμβολιασμό, μου είπαν ότι τα εργαστήρια είναι υπεύθυνα μόνο για την ποιότητα των εμβολίων ο οργανισμός φαρμάκων θα δώσει την έγκριση και μετά τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για την χρήση. Οπότε ρωτάω εγώ, αν εγώ εμβολιαστώ και έχω μία ασθένεια νευρολογική, την Κιγέμ Μπαρέ, σε ποιον θα πάω να απευθυνθώ, στην κυβέρνησή μου, στον ΕΜΕΑ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Στις Ηνωμένε Πολιτείε τα εργαστήρια απέκτησαν οι φαρμακοβιομηχανίες απέκτησαν ασυλία. Δεν θέλω να δω το ίδιο πράγμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να αναφέρω. Αυτό που έγινε στην Baxter. Η Baxter πέρυσι χρησιμοποίησαν ένα εμβόλιο που οδήγησε στο θάνατο πολίτες της Τσεχοσλοβακίας και το ίδιο συνέβη και στην Αυστρία και υπήρξε και σχετική δίκη. Το ερώτημα που θέλω να θέσω λοιπόν στην Επίτροπο είναι πόσο αξιόπιστα μπορεί να είναι τα πρωτόκολλα ασφαλείας των φαρμακοβιομηχανιών και τι θα κάνετε προκειμένου τα πρωτόκολλα φαρμακοεπαγρύπνησης να χρησιμοποιούν ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα παρακολουθούν και τον εμβολιασμό και τα εμβόλια προκειμένου να διαπιστώσουμε ότι η όλη διαδικασία είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από τις βιομηχανίες. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να... Και ελπίζω να θυμάμαι όλα αυτά που με ρωτήσατε. Λοιπόν, το κατά πόσο το εμβόλιο είναι ασφαλές για τα παιδιά και τις αγγείους. Φυσικά, στη συνέχεια, ο εμπειρογνώμονας θα μπορέσει να σας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα πιο συγκεκριμένα. Να σας πω τι γνωρίζω εγώ για το θέμα. Γνωρίζω ότι ο Οργανισμός για τα Φάρμακα, όταν δημοσίευσε ε, τη δική του επιστημονική γνωμοδότηση, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρεί κανείς ότι αυτό το εμβόλιο είναι μη ασφαλές για τα παιδιά και τις εγγύους. Μέχρι σήμερα έκαναν 9.000 κλινικές δοκιμές και ζήτησαν επίσης από τις ενδιαφερόμενες φαρμακευτικές εταιρείες να συνεχίσουν τις δικές τους κλινικές δοκιμές για τουλάχιστον ε, άλλες 28.000 ε, περιπτώσεις, δίνοντας έμφαση στα παιδιά και στους Πιστεύουν ότι επειδή το δίπλωμα ευρεσιτεχνία για την παραγωγή εμβολίου ε, είναι το ίδιο για την γρήπη τα τελευταία 20 χρόνια, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρούν ότι δεν θα συμπεριφερθεί διαφορετικά το εμβόλιο αυτό από, σε σχέση με τα προηγούμενα. the... Αλλά βεβαίω η οδηγία για τη φαρμακοεπαγρύπνηση της, του οργανισμού για τα φάρμακα είναι πολύ αυστηρή σε αυτήν την περίπτωση. και όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Δηλαδή, η αρμόδια ε, για την άδεια, ε, αρμόδιος φορέας για την άδεια στα κρατημέλη κτλ. Όλοι έχουν καθήκον να αναφέρουν την παραμικρή παρενέργεια που θα υποπέσει την αντίληψή τους. Και ο τα Φάρμακα αλλά και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη των, ε, νότων Νόσων θα, θα παρακολουθήσουν την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή. Έτσι ώστε στην περίπτωση που υπάρξει ε, κάποια απόδειξη για ε, ανεπιθύμητες ενέργειες, τότε ο Οργανισμός για τα Φάρμακα θα ε, αλλάξει την γνωμοδότησή του. Και βεβαίως αυτό θα επηρεάσει κατάλληλα και την διαδικασία έγκρισης, εάν χρειάζεται βέβαια. Εποχιακή γρήπη. Η εποχιακή γρήπη βεβαίως και είναι σοβαρή και δεν νομίζω ότι θα συμφωνούσα με οποιοδήποτε που θα ισχυριζόταν το αντίθετο. Όταν, όπως σας είπα, ε, από ε, 200, ε, θύματα το χρόνο έχουμε. δεν πρέπει να υποτιμάμε τη σοβαρότητα ακόμα και της εποχιακής γρήπης. ούτε και αυτή. Παρόλο που ε, τα ποσοστά θνησιμότητα είναι παρόμοια με τα ποσοστά θνησιμότητα τη εποχιακή γρήπη. Ε, πώ τώρα δίνουμε τι πληροφορίε στο κοινό, πώ επικοινωνούμε το κοινό. Ναι, συμφωνώ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και στη νέα μα ανακοίνωση, στο έγγραφο εργασία που, που αναφερόμαστε στην ε, επικοινωνία με το κοινό, λέμε ότι στι 12 Οκτωβρίου θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τους Υπουργού Υγεία θα προτείνουμε να αποφασίσουμε μία συγκεκριμένη μέρα, να ε, πούμε τα ίδια πράγματα και στα 27 κράτη-μέλη. Συμβουλές προς το κοινό, για το βόλιο, για τα πάντα. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε την ομοιόμορφη παροχή πληροφοριών προς το κοινό. Με την προϋπόθεση βέβαια θα συμφωνήσουν και οι υπουργοί και θα δεχτούν τις συμβουλές αυτές. Well, I think this is all. Okay. Merci beaucoup. Εντάξει, λέει ο ε, ο Τόμας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ και την κυρία Επίτροπο για την παρουσία της και για τον θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει η Κομισιόν και ελπίζω ότι θα μπορέσω να έχω νέα στοιχεία από αυτά που θα μας πει για τα θέματα της ε, των παρενεργειών. Σίγουρα όταν εμβολιάζουμε ένα εκατομμύριο ασθενείς κάποιες παρενέργειες θα επανέλθουν, θα εμφανιστούν. Η, η γερμανική νομοθεσία λέει ότι στην ε, περίπτωση των ε, ρυθμίζει τα θέματα της αστικής ευθύνης για την περίπτωση παρενεργειών. Επίσης, επειδή υπάρχουν, ε, υπάρχει παρουσία μετάλλων στα εμβόλια αυτά, θα ήταν χρήσιμο να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση φαρμάκων τα οποία δεν περιέχουν σε επίπεδο ιχνών μετάλλια, με, μέταλλα. Και χωρίς αυτό να τροποποιήσει το, την αντιγόνο δράση των ε, εμβολίων αυτών. Νομίζω επίση για την εκστρατεία πληροφόρηση, νομίζω ότι η Κομισιόν μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της, να έχει παραγματικά χάρη μηνύματα συνθηματολογικού χαρακτήρα όπως πλένετε τα χέρια σας κάθε μέρα, τα οποία μπορεί να είναι απλές ε, προσκλήσεις προς τον πληθυσμό που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν οι πολίτες. Ένα ακόμα ερώτημα στην Βουλγαρία υπάρχουν πολλοί συνοριακοί σταθμοί όπου ο καθένας που μπαίνει στην ε, ε, Βουλγαρία ή βγαίνει από τη Βουλγαρία πρέπει να παρουσιάσει ένα πιστοποιητικό για το γεγονός ότι δεν έχει ε, την γρήπη αυτή. Αλλιώς πρέπει να πληρώσει 80 ευρώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι του οποίου πρέπει να επιληφθεί η Κομισιόν. Επόμενος ομιλητής η Αντώνια Παρβάνουα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Με εντυπωσιάζει ιδιαίτερα η προσέγγιση σας, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε μια συγκεκριμένη επιδημία ή πανδημία γρήπη στην Επιτροπή μας. Η πρώτη, αφορούσε, η πρώτη φορά το θέμα ήταν η γρήπη των πτηνών, τώρα έχουμε τη γρήπη των χείρων, ελπίζω να μην έχουμε την γρήπη των ψαριών. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί ως τα δυνατόν ε, να ακολουθήσει μια πρακτική προσέγγιση. Είναι προφανές από αυτά που μας είπατε ότι δεν υπάρχει ε, αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε σχέση με την εποχιακή γρήπη. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Και ταυτόχρονα προτείνεται ένα ευρύ φάσμα μέτρων για τον συντονισμό και την συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ναι, αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και αυτή θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι ο βασικό ρόλο τη Επιτροπή είναι η εκπαίδευση. Κοιτάξτε, στο 21ο αιώνα δεν νομίζω ότι ο ρόλο τη Επιτροπή είναι να λέει στου ανθρώπου ότι πρέπει να πλένονται και να παίρνουν τα χέρια του. Αλλά ρωτώ το εξή. Εσεί αισθάνεστε εμπιστοσύνη όσον αφορά τα εμβόλια και ε, το κίνδυνο. Μιλώ γιατί εδώ μιλάμε για επιταχυνόμενες διαδικασίες έγκρισης και μήπως θα πρέπει να, να ενταθεί η φαρμακοεπαγρύπνηση γιατί... για τις παρενέργειες. Γιατί αν θέλετε αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θα θέσουν και οι πολίτες. Όσον αφορά τις εγγύους και τα παιδιά ε, με άσθημα, Κοιτάξτε, ε, μιλάμε για κατηγορίες που συνήθως ε, δεν πρέπει να εμβολιάζονται. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι με τα προβλήματα υγείας επηρεάζονται και παρουσιάζουν την υψηλότερη, τα υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητα. Από την έχουμε αυτό και από την άλλη το γεγονός ότι αυτού του ανθρώπου ακριβώ δεν του εμβολιάζουμε συνήθω. Άρα λοιπόν ρωτώ, τι πρέπει να κάνουμε. Μήπω πρέπει να κάνουμε ε, υπηρεσίε συνειδητοποίηση και ενημέρωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαδώσει αυτέ τι πληροφορίε ε, στα κράτη-μέλη. Να ξέρουμε ποιο είναι ο βαθμό επιπολασμού και τι γίνεται με τον βαθμό νοσηρότητα. Well, ε, Κοιτάξτε. Όπως δεν απαντήσατε για το θέμα της Βουλγαρίας, θα απαντήσω εγώ. Με πληροφορούν οι υπηρεσίες ότι έχουν θέσει αυτό το ερώτημα των ε, πιστοποιητικών στα σύνορα που ζητείται πιστοποιητικό ότι κανείς δεν έχει την ε, γρήπη αυτή και από ό,τι γνωρίζουν δεν είναι επίσημη πολιτική της βουλγαρικής κυβέρνησης, είναι απλώς κάποιοι συνοριακοί φύλακες οι οποίοι έχουν πάρει αυτή την πρωτοβουλία <laughs> να κάνουν αυτές τις ερωτήσεις για το αν υπάρχουν ή όχι πιστοποιητικά. Τώρα, το ερώτημά σας, αν πράγματι εμπιστεύομαι τα εμβόλια αυτά σε ό,τι αφορά το, την ασφάλεια. Εγώ μπορώ να πω μονάχα ότι εμπιστεύομαι τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αλλιώς θα είχαμε τέτοιους επιστημονικούς φορείς που μας αρρωγούν και μας συμβουλεύουν. Έχω εμπιστοσύνη στον Οργανισμό Φαρμάκων και στον Οργανισμό για την Πρόληψη των Ασθενειών. Όταν μου λένε ότι αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές, τους έχω εμπιστοσύνη. Αυτό το οποίο λένε λοιπόν οι φορείς είναι ότι γνωρίζοντας τις συνέπειες που μπορούν να προκύψουν για ένα άτομο το οποίο έχει ήδη προβλήματα υγείας εάν δεν τύχει εμβολιασμού, αν κάνει κανείς μία ανάλυση κινδύνου σε σχέση με όφελος, το όφελος φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο από τον κίνδυνο. Σε τελική ανάλυση τελικά είναι ο θεραπονίατρος ο οποίος πρέπει να συμβουλεύσει ένα άτομο αν πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι. Αλλά οι συμβουλές του Οργανισμού Φαρμάκων είναι ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση το κέρδος είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο. Ε, παρέλειψα να απαντήσω <clears throat> σε ένα ερώτημα για το θέμα της αστικής ευθύνης σε περίπτωση παρενεργειών για τα φάρμακα. Καταρχήν είναι ο παραγωγός των φαρμάκων. Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο οργανισμός παράγει το φάρμακο, η εταιρεία παράγει το φάρμακο, έχει την ευθύνη. Δεύτερον, είναι ο θεράπον, ο ιατρός ο οποίος δίνει τη συμβουλή για τον εμβολιασμό και φυσικά και η εθνική κυβέρνηση η οποία έχει εγκρίνει ένα συγκεκριμένο φάρμακο για την θέση του σε εμπορία. Έχουμε λοιπόν τρία επίπεδα αστικής ευθύνης στην περίπτωση παρενεργειών. Για τα εμβόλια τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν καθόλου ίχνη μετάλλων, φοβάμαι δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το ερώτημα, ενδεχομένω μπορείτε να το θέσετε στον ε, Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Φαρμάκων. Ο Φίλιπ Σουβά τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ορισμένε ερωτήσεις. Καταρχάς, είπατε ότι η θνησιμότητα της ε, γρήπης δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή της ε, εποχικής γρήπης. Αυτό το σημειώνω με ενδιαφέρον γιατί αρκετές επιστημονικές δημοσιεύσεις ε, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο έδιναν άλλα νούμερα. Ορισμένε μάλιστα έλεγαν ότι η θνησιμότητα θα μπορούσε να είναι μέχρι και τέσσερι φορές μεγαλύτερη από αυτή της εποχιακής γρήπη. Αυτό το θέμα είναι σημαντικό γιατί βεβαίως μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό θανάτων αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία. Είναι αλήθεια βεβαίως ότι τα επιστημονικά δεδομένα εξελίσσονται συνεχώς και ότι τα δεδομένα του Ιουνίου και του Ιουλίου δεν είναι τα ίδια που θα έχουμε τον Οκτώβριο, γιατί προσαρμόζεται και η επιστημονική κοινότητα στα δεδομένα. Όμως, θεωρείτε ότι οι επιστήμονες πέρασαν από μία εκτίμηση που μιλούσε για τετραπλάσια θνησιμότητα σε μία εκτίμηση που μιλάει για ίση θνησιμότητα με την επιφυσιακή γρήπη. Δεύτερο ερώτημα, όσον αφορά τις παρενέργειες των εμβολίων. Είναι αλήθεια ότι για όλα τα φάρμακα υπάρχουν παρενέργειες. Το ερώτημα είναι, η σχέση ωφέλειας κινδύνου είναι υπέρ μας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Παρενέργειες πάντα υπάρχουν. την περίπτωση της εποχικής γρήπης μιλάμε για ένα στο ένα εκατομμύριο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το ίδιο κίνδυνο. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο στατιστικά να μιλήσουμε για μη ύπαρξη παρενεργειών. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι υποθέσεις όμως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι η σχέση κινδύνου ωφέλειας. Και να πω ότι αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αγοράσει εμβόλια, ορισμένες φορές σε μαζικές ποσότητες. Θα ήθελα όμως να μου πείτε γενικά σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά εμβολίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θεωρείτε ότι είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι και από εκεί και πέρα πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια ισότιμη μεταχείριση. Γιατί όπως είπατε και εσείς υπάρχουν και οι χώρες ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που χρειάζονται εμβόλια. Εγώ σας ρωτώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνετε προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στα εμβόλια από όλους με βάση την εθνική πολιτική. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σταταρέλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, την κυρία Επίτροπο γιατί ήρθε σήμερα εδώ για να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων και σας ευχαριστούμε για τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε για το που βρισκόμαστε και για τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν ή που πρόκειται να εγκριθούν ε, για να συγκρατήσουμε ε, την ε, πανδημία της γρήπης ΝΙΑΝΑΙΤΑΕΝΑ. Κοιτάξτε, από την παρουσίασή σας νομίζω ότι κατάλαβα ότι πιστεύετε ότι η κατάσταση είναι κάτω από έλεγχο. Τώρα, Χωρί αυτό σημείο δεν αποκλείουμε ε, την επιδείνωση τη κατάσταση. Τα τελευταία δέκα χρόνια πρέπει να πω ότι είχαμε ξέσπασμα τη ε, γρήπη των πτηνών, το SARS και τώρα την, ε, αυτή τη συγκεκριμένη επιδημία γρήπης και όλα αυτά έχουν αποδείξει το πόσο ορισμένες ζωονόσοι μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο και το αντίστροφο. Δηλαδή, ε, ε, να μολύνθηκε ο άνθρωπος και στη συνέχεια με τη σειρά του ε, να μόλυνε τα ζώα. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να δούμε ότι στο μέτωπο της πρόληψης δεν έχουμε ακόμα τα κατάλληλα μέσα για να αποφύγουμε δραματικές απώλειες και ανθρωπίνων ζώων αλλά και αποδεκατισμό των ζώων. Μήπως λοιπόν έφτασε η στιγμή, δεν θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα αποτελεσματικό ολοκληρωμένο σύστημα επαγρύπνησης των ζωονόσων που να συνδυάζει τον τομέα της ανθρώπινης υγείας και τον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας. Όπως, το, όπως γνωρίζετε, ε, το να αντιμετωπίσουμε τις επίγουσες καταστάσεις κοστίζει πολύ και τα στοιχεία που έχουμε είναι εντυπωσιακά. το 65% ε, των λιμωδών νόσων ε, που ξέσπασαν τα τελευταία 60 χρόνια προήλθαν από ε, παθογένειες που μεταπίδησαν από το ένα είδος στο άλλο. Τα τελευταία 10 χρόνια οι απώλειες οικονομικές ξεπερνούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα 140 δις ευρώ. Άρα, σε κάθε επίγουσα κατάσταση, και τα ξέρουμε όλα, ε, τι έχουμε, ε, ε, παρεμπόδιση των εμπορικών συναλλαγών, ε, προειδοποίηση των ταξιδιωτών, ε, ε ομαδικές σφαγές χιλιάδων ζώων, ε, τροποποίηση των, της διατροφής μας, αποκλείοντας ορισμένα είδη από τη διατροφή μας. Δεν συνέβη και με τα, τα πουλερικά, δεν συνέβη και με τις αγελάδες, τώρα συνέβη και με τους χείρους. Σα ρωτώ λοιπόν, δεν ήρθε η στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε μία λύση που να προωθεί μόνιμη συνεργασία ανάμεσα στην ιατρική και στην κτηνιατρική έτσι ώστε να έχουμε ε, ε, λειτουργικό, ένα ολοκληρωμένο, αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα ελέγχου που να καλύπτει όλε τι πτυχέ ε, τη ανθρώπινη υγεία. Και από την παραγωγή μέχρι την πώληση των ειδών διατροφή. Πρώτον, σύστημα συνολική επαγρύπνηση και παρακολούθηση που θα βλέπουμε αμέσω το που δημιουργούνται νέα στελέχη που μεταπηδούν από τα ζώα στου ανθρώπου και το αντίστροφο. Δεύτερον, πρόθεση συνολικών μέτρων προληπτικών για του εργαζόμενου σε ορισμένου Τρίτον, καθορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο του επίπεδου βιοασφάλεια για να περιορίσουμε τη μετάδοση των ιών ε, στα, στα ζώα. Ε, ε, ε Επίση, ε, να μπορούμε να συλλέγουμε αξιόπιστα στοιχεία, να τα διαχειριζόμαστε και να τα δίνουμε σε όλε τι γωνιέ τη γη. Επίση, ενίσχυση τη συνεργασία ανάμεσα στα κέντρα αριστεία που ασχολούνται με θέματα ιατρική και κτηνιατρική και τέλο να δημιουργήσουμε ένα μια πολυτομιακή τεχνική ομάδα που να είναι ικανή να επεξεργαστεί σωστέ ομάδε, σωστέ ε, προτάσει, συγγνώμη, για τη σωστή διαχείριση του συστήματο. Με δύο λόγια. Δεν ήρθε η στιγμή να δούμε γενικά και σε προληπτικό επίπεδο αυτά τα προβλήματα, αντί να τρέχουμε διαρκώ όταν ε, προκύπτουν αυτέ οι επίγουσε καταστάσει. Ευχαριστώ. Ήταν μακροσχελής η κατάληξή σας, αλλά ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει σήμερα το απόγευμα. Νομίζω και εγώ ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πρέπει να αλλάζει ρούχα και να πλένεται. Νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσουμε όμως σε όλους ότι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους πιο συχνά. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της ε, συναδέλφου μας της Dagmar Roth Berend είδα κάποιους διερμηνείς να απολυμμένουν τα χέρια τους με τα ειδικά μαντιλάκια. Ή μάλλον το κάναν και πάλι όταν λέγαμε για την ανάγκη της καθαριότητας και της ανάγκης να χρησιμοποιούμε αυτά τα μαντιλάκια καμιά φορά. Νομίζω λοιπόν ότι οι σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες είναι πάντα επωφελείς. Εγώ μίλησα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας στη Ρουμανία σε σχέση με την κατάσταση στην ε, Ρουμανία και ρώτησα τον αρμόδιο υπουργό ποιες περιοχές είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο. Μου είπε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι όταν ταξιδεύετε σε ένα αεροπλάνο ή περνάτε από αεροδρόμια. Έχετε να προτείνετε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τα αεροδρόμια και τα αεροπλάνα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλα τα μέτρα είναι γενικά μέτρα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να απαντήσω εδώ στα ερωτήματα αυτά. Καταρχήν, για τη θνησιμότητα, για το ποσοστό θνησιμότητος. Δεν ξέρω αυτό το οποίο λέτε για το ότι η ΙΤΑ 1 1 έχει τετραπλάσια θνησιμότητα από την εποχική γρήπη. Δεν ξέρω από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία. Είπατε ότι το είδατε κάπου να έχει δημοσιευτεί τον Ιούνιο. Βάσει αυτών που γνωρίζω εγώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μην λησμονήσετε και το είπατε και ο ίδιος σας ότι οι πληροφορίες είναι ρευστέ, ότι αλλάζουν συνέχεια. Τώρα έχουμε τουλάχιστον συλλέξει την εμπειρία του νοτίου ημισφαίριου από το οποίο παίρνουμε σε καθημερινή βάση τις πληροφορίες και παρακολουθούμε σε καθημερινό επίπεδο <clears throat> ποια, πόσα είναι τα περιστατικά που παρουσιάζονται και ποια είναι η θνησιμότητα. Βάσει των πληροφοριών που έχουμε, η θνησιμότητα φαίνεται να είναι ακριβώς η ίδια όπως και στην εποχική γρήπη. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο μέλλον, προ το παρόν όμω ούτω έχουν τα πράγματα. Συμφωνώ τώρα μαζί σα ώστε για να μπορέσουμε να κρίνουμε το αν θα πρέπει κανείς να εμβολιάζεται ή όχι, αυτό σε τελική ανάλυση είναι προσωπική επιλογή του κάθε ατόμου, φυσικά σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό. Και πρέπει κανείς να ζυγίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους και την ωφέλεια. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να καταλήξει κανείς σε μια απόφαση. Θέσατε και ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σε σχέση με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη από την αρχή θυμάμαι ότι κατά τη διάρκεια ακόμα της Γαλλικής Προεδρίας εμείς είχαμε συζητήσει το θέμα του να δημιουργήσουμε ένα αποθεματικό εμβολίων σε ευρωπαϊκή βάση από το οποίο όλα τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να αντλούν εμβόλια. Τα κράτη-μέλη είπαν όλα όχι, θέλουμε να έχουμε τα εθνικά μας αποθέματα δεν τους άρεσε η ιδέα του να υπάρχει ένα τέτοιο αποθεματικό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν ο κάθε υπουργό να αποφασίσει τι είναι απαραίτητο για τη δική του χώρα, πόσα εμβόλια είναι απαραίτητο να έχουν προμηθευτεί και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολυπικιλία αντιμετωπίσεων μεταξύ των κρατών μερών. Υπήρξαν χώρες που παραγγείλαν εμβόλια για όλο τον πληθυσμό τους, άλλες για το μισό του πληθυσμού τους, άλλες χώρες για 20% του πληθυσμού τους. Και έχουμε ακόμα και κράτη-μέλη που δεν έχουν αγοράσει καθόλου εμβόλια. Θα επιτρέψουμε λοιπόν στα κράτη-μέλη αυτά να εκτεθούν σε μία υγειονομική απειλή. Σίγουρα όχι. Αυτό στο οποίο εγώ προσπαθώ είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε μια καλύτερη μορφή συντονισμού και αρρωγής προς τα κράτη-μέλη αυτά ώστε να έχουν μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού βάσει της οποίας θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εμβόλια. Και αυτή τη στιγμή εμείς αναπτύσσουμε μια διαδικασία υποβολής ε, προσκλήσεων σε, για ένα δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια εμπορίων, εμβολίων για 10 κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη που έχουν παραγγείλει πάρα πολλά εμβόλια περιμένοντας τη γνωμοδότηση αυτή που θα πει ενδεχομένω ότι μία δόση του εμβολίου ενδεχομένω θα επαρκεί, ενώ η αρχική γνωμοδότηση έλεγε ότι δύο χρειάζονται, στι ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μία δόση είναι, είναι αρκετή, γιατί δεν χρησιμοποιούν προσθετικές ουσίες. Ίσως στο μέλλον θα αναθεωρήσουμε και εμείς την απόφαση αυτή, γιατί, λέ... γιατί ενδεχομένως να φτάνει μία δόση μονάχα και να μην χρειάζονται δύο. Οι χώρε αυτές λοιπόν που έχουν προμηθευτεί πάρα πολλά εμβόλια γιατί βασιζόντουσαν στο ότι χρειάζονται δύο δόσεις, λένε τώρα ότι μπορούν να ξαναπουλήσουν, να μεταπολίσουν μερικά από τα εμβόλια τους σε άλλες χώρες. Επομένως, συμμετέχουν στην προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν και για τα υπόλοιπα 10 κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί εμβόλια να υπάρχουν οι απαραίτητε δόσει. Το ερώτημα τώρα της ε, μόλυνσης από τα ζώα. Έχουμε χειροτροφία, τα οποία είχαν πληγεί από τον ιό του ΙΤΑ 1 νι 1 στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αργεντινή και τώρα και στην Βορειοελλανδία. Τρία χειροτροφία στη Βορειοελλανδία έχουν πληγεί από αυτό τον ιό. <clears throat> Αλλά έχουμε ένα, μια κοινή δήλωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τον ΦΑΟ και από άλλους φορείς λέγοντας ότι ο ιός ή τα ένα ή ένα δεν μπορεί να περάσει από το ένα είδος, από τους χείρους στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει σύμφωνα με αυτές τις εμπειρογνωμοσύνες. Και γι' αυτό πήγα εγώ πρόσφατα στην Κίνα και έθεσα αυτό το ερώτημα στις κινέζικες αρχές. Γιατί οι κινέζικες αρχές εξετάζανε τη δυνατότητα να κάνουν κάποιους περιορισμούς για την εισαγωγή χοιρινού κρέατος από ορισμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τους θα πρέπει να παραμείνουν στο επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων τους, είναι μέλη και των τριών αυτών διεθνών οργανισμών που έκαναν τη δήλωση που προανέφερε, επομένως θα πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Και μου υπεσχέθηκαν ότι θα αναθεωρήσουν την απόφασή τους. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ότι θα μειώσουν τους περιορισμούς και θα αναθεωρήσουν ενδεχομένω και πλήρω την απόφασή του. Για το θέμα τώρα της ε, μόλυνσης ανθρώπων και ζώων από τη γρήπη στις 30 του επομένου μηνός οργανώνουμε μια σημαντική διάσκεψη που έχει σαν τίτλο «Μία και μοναδική είναι η υγεία» και όπου θα είναι η αρχικτινία τρίτων κρατών μελών και η αρχή των κρατών μελών για να συζητήσουν τη σχέση μεταξύ ζωικής υγείας και ανθρώπινης υγείας και διασταυρουμένων μολύνσεων μεταξύ ζώων και ανθρώπων. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν συνδιάσκεψη. Αν σας ενδιαφέρει θα μπορούσα να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την ε, συνδιάσκεψη. Ο κύριος Λάνιου έχει το λόγο. Κυρία Λάνιου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι στους ε, αγγλόφωνους ε, συναδέλφους και σας λέω το εξής μην χρησιμοποιούμε άλλο τον όρο swine flu, γιατί αυτό κάνει το BBC. Αυτό ακούμε στα, στα αγγλικά διαρκώ. Γρήπη των χείρων. Καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα με του χειροτρόφου μα, διότι η Κίνα βρίσκει πρόσχημα και στα αγγλικά και στον αγγλικό τύπο. Ε, μην το συνδέετε με τη γρήπη των χείρων, γιατί δεν υπάρχει αποπιστημονική ε, από άποψη, δεν ευσταθεί αυτή η συσχέτιση. Τώρα, για τι ομάδε κινδύνου. Έχω την εξαιρώτηση. Αναφέρετε στην ανακοίνωσή σα ότι. Ε, ε, υπάρχει μία κατηγορία πρώτον το ε, ιατρικό προσωπικό. Ε, αντίθετα με το τι γίνεται στις Ηνωμένε Πολιτείε, Νέα Υόρκη και αλλού, εδώ σε εμά, εάν είναι κανεί μέλο ιατρικού προσωπικού, ιατρό ή μέλο νοσηλευτικού προσωπικού, έχει το δικαίωμα επιλογής. Στη χώρα μου δεν βλέπω και τρομερό ενθουσιασμό, δεν στριμώχνονται όλοι και από ό,τι μου αναφέρουν Δεν κρατούν καν ε, αρχεία τα νοσοκομεία για το ποιο εμβολιάστηκε και ποιο όχι. Αν, επεκταθεί όμω ε, ε, η επιδημία, θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε ποιο εμβολιάστηκε ή όχι. Στα πλαίσια επίση εθνική στρατηγική θα χρειαζόμαστε τα στοιχεία. Να κλείσουμε τα σχολεία, από την άλλη όμω, ε, να, ε, καταλαβαίνετε κάποιος θα πει ότι ζητήστε από, από τον, τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού που δεν έχουν εμβολιαστεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά. Καταλαβαίνετε τι πρόβλημα θα δημιουργήσει αυτό, Κυρίω θα μιλάμε για κράτη-μέλη που έχουν και λίγου γιατρού και ε, λίγους νοσηλευτές. Πώς θα ε, παροτρύνετε λοιπόν τα κράτη-μέλη για να εμβολιάσουν αυτέ τι ομάδε. Επίση, οι έγκυε γυναίκε. Ε, το θέμα φαίνεται ότι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είπατε και οι ίδιοι στα αγγλικά ε, ότι δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι ότι είναι ε, επικίνδυνο το εμβόλιο. Εγώ νομίζω όμως ότι τα κράτη-μέλη βλέπουν τελείως διαφορετικό το θέμα όταν αρχίζουν να μιλούν για τις διάφορες ομάδες κινδύνου. Στην ε, χώρα μου λένε για παράδειγμα προ Θεού κανένα εμβολιασμό κατά τη διάρκεια του πρώτου τρει μήνε τη κοίηση. Σε άλλε χώρε λένε όχι, αυτό είναι το ιδανικό χρονικό διάστημα γιατί εκεί ε, είναι, ε, ε, το, το, το, το όφελο είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβόλιο από το κόστο. Το ίδιο και όσον αφορά τα NDAK, τα μυφλού και άλλα. Ε, ε, ε, αντιφατικά στοιχεία. Για παράδειγμα, τι γίνεται, ε, με, πώς επιδρούν τα φάρμακα αυτά στο έμβριο Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι το θέμα αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ε, όσον αφορά δηλαδή τις συνέπειες στο έμβριο. Μιλώ συγκεκριμένα για τη λήψη αντιοικών από την έγκυο μητέρα. Και τέλο πάντων, οι τεχνικέ πληροφορίε ε, θα τι ακούμε, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Εμένα με νοιάζει η, η σαφήνεια. Γιατί ωραία όλα αυτά. Επικουρικότητα, ρίχνω το, στέλνω τον μπαλάκι στα κράτη-μέλη. Αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να ακολουθήσει μία και μόνο εδώ. Και ε, οι πολίτε είναι ευφυεί. εκεί κοιτούν και τι κάνουν οι γείτονε. Αν ε, ακούσει λοιπόν ο πολίτη στι κάτω χώρε, για παράδειγμα, του τρει πρώτου μήνε τη κοίηση, ε, αποθαρρύνει τον εμβολιασμό ε, και στη Γερμανία γίνεται ακριβώ το αντίστροφο, τότε καταλαβαίνετε ο πολίτη αρχίσει να έχει ε, αμφιβολίε, θα πει Α, εδώ έχουμε αντιφατικέ πληροφορίε, δεν κάνω τίποτα, δεν εμβολιάζομαι. Επίση, κάτι άλλο. Είπατε την ίδια μέρα να βαθεί το ίδιο μήνυμα παντού στην Ευρώπη. Μα κοιτάξτε, σήμερα ε, τόσο, ακούμε τόσο αντικρουόμενα μηνύματα μεταξύ του, που ε, τελικά ο πολίτη δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και θα πει δεν εμβολιάζομαι καθόλου. Τι, πώ θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Δύο ακόμα παρεμβάσει. Ο Ρίχα Τσέμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα απλό ερώτημα για την κυρία Επίτροπο. Υπάρχουν ε, διάφορες, ε, διάφορα σκευάσματα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια είναι η αποτελεσματικότητα, ποια είναι η δραστικότητα αυτών των ουσιών. Και επίσης υπάρχουν ε, ορισμένες ε, συγκρίσεις αυτών των σκευασμάτων με γενετικού χαρακτήρα ε, φάρμακα αντιϊκά. Πώς εκτιμάτε λοιπόν αυτήν την ε, διαφορά. Επίσης, μήπως έχει η Κομισιόν κάποιες ε, αρμοδιότητες στον τομέα αυτό της υγείας να προχωρήσει και σε μια πληροφοριακή εκστρατεία προς τον πληθυσμό για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να προωθήσει κάποια πολύ απλά μηνύματα με τα οποία μπορεί να υπάρξει κάποια προς κάποια πρόληψη. Πιστεύω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το εμποδίσει να κάτω μέλος αν εσείς το θεωρείτε αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση σε σχέση με τις απαντήσεις σας. Είπατε ότι εμπιστεύεστε την ΕΜΕΑ. Ναι, Όντως, αλλά ο ρόλος σας είναι διαφορετικός από τη ΣΕΜΕΑ. Ο ρόλος της ΕΜΕΑ είναι να αναλύσει τους κινδύνους και τις ωφέλειες για ένα στέλεχος. Η δική σας δουλειά είναι να δείτε τι συνέπειες θα υπάρξουν για άλλες ε, ευρωπαϊκές ε, νομοθεσίες. Για παράδειγμα, περιέχουν υδράργυρο, υπάρχουν άλλες μέθοδοι που είναι περισσότερο οικονομική και λογική από οικονομικής φύσης. Οπότε είναι διαφορετικός ο ρόλος σας και δεν αρκείτε στο να σφραγίσετε κάτι. Το ίδιο ισχύει και για το τρόφιμα ας πούμε. Η ΕΦΣΑ μπορεί να αποφασίσει για την έγκριση όχι κάποιου προσθέτου, αλλά εσείς έχετε διαφορετικά κριτήρια. Πρέπει λοιπόν να κάνετε διάκριση μεταξύ ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης κινδύνου. Διαχείριση κινδύνου είναι ο δικός σας ρόλος και πρέπει να υπάρξει διάκριση. Let Ας ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση. Εμπιστεύομαι την ΕΜΕΑ και τον ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών, γιατί γνωρίζω ότι κάνουν πλήρη εκτίμηση και διαθέτουν τις υποδομές και τις πληροφορίες που χρειάζονται για να κάνουν μία ολοκληρωμένη εκτίμηση των συνοποιών οποιοδήποτε φαρμάκου. Και γι' αυτό συστήσαμε αυτούς τους οργανισμούς. Όχι για να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, αλλά γιατί χρειαζόμασταν επιστημονική στήριξη για να λαμβάνουμε αποφάσεις και θα σας πει και η ΕΜΕΑ ότι έχει κάνει μελέτες και για θέματα όπως την παρουσία υδραργύρου. Δεν γνωρίζω εγώ τις λεπτομέρειες, αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορούν να σας απαντήσουν στο θέμα αυτό. Βεβαίως, είναι καθήκον μας να παρακολουθούμε τα πάντα και να είμαστε προετοιμασμένοι να αλλάξουμε τη στάση μας οποιαδήποτε στιγμή αν θεωρούμε ότι συνάδει τέτοιος λόγος, αν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Τώρα, για το κατά πόσο ο εμβολιασμός πρέπει να είναι προαιρετικός ή όχι. Θεωρώ ότι ο εμβολιασμός είναι επιλογή του κάθε ατόμου. Βεβαίως, είναι υποχρέωσή μας να δώσουμε συμβουλές και θα δώσουμε συμβουλές με βάση όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει. Όμως δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τους γιατρούς να εμβολιαστούν αν δεν το επιθυμούν. Όπως είπα και πριν, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις ομάδες επικινδυνότητας. Και αυτές οι ομάδες είναι οι ίδιες που αναφέρει και ο ΠΟΗ. Άτομα που ήδη έχουν προβλήματα υγείας έγκυες γυναίκες και άτομα που εργάζονται στον τομέα της υγείας. Οπότε, η δική μας συμβουλή είναι ότι οι γιατροί και οι νοσοκόμες πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Βεβαίως, αν δεν το επιθυμούν, δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε. Τώρα, καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε ότι στέλνω διαφορετικά μηνύματα. Όμως, αυτό δεν το κάνουν μόνο οι Υπουργοί. Πολλοί στέλνουν αντικροούμενα μνήματα. Κάθε μέρα μαθαίνω ότι έγινε μία έρευνα στην τάδε χώρα που δείχνει αυτό. Έγινε άλλη έρευνα σε άλλη χώρα που δείχνει κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά όταν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα στον πληθυσμό και προκαλούν σύγχυση. Όμως υπάρχουν και οι επαγγελματίες. Και επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε επιστημονικούς οργανισμούς που συλλέγουν όλες τις πληροφορίες, όλες τις έρευνες και δημοσιεύουν τις γνωμοδοτήσεις τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε προσέξει πάρα πολύ το θέμα της ενημέρωσης του κοινού και θα το συζητήσουμε και με τους Υπουργούς Υγείας τον Οκτώβριο και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε να υπάρξει ένα κοινό ανακοινοθέν για τα 27 κράτη-μέλη που θα περιλαμβάνει τα βασικά σημεία τουλάχιστον. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε για τις ε, απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα που ετέθησαν. Θεωρώ ότι όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες προετοιμασίας και οργάνωσης και να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχουν οι δυνατότητες εμβολιασμού και θα δούμε τι θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου όταν θα γίνει η επόμενη συνάντηση των Υπουργών ε, Δημόσιας Υγείας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή η πληροφόρηση προς την κοινή γνώμη θα κάνει απλούστερη την αντιμετώπιση και θα βοηθήσει και τα κάτι μελη να δώσουν πιο στοχευμένες πληροφορίες προς την κοινή γνώμη. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας, λέει η κυρία Βασιλείου. Μπορούμε να συνεχίσουμε την ε, ημερήσια διαταξή μα. Έχουμε τώρα τη συζήτηση με τον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Φαρμάκων, τον κύριο Τόμας Λέντγκρεν. Αν θέλετε να έρθετε στο, έδρανο των στο προεδρικό έδρανο, κύριε Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε την ημερήσια διάταξη. Χαιρετίζω την παρουσία του κ. Τόμα Λίντγκεν, ο οποίο είναι εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού Φαρμάκων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλώ ήλθατε. Έχετε μαζί σα τον κύριο Μάρκο Καβαλιέρη, ο οποίο είναι εμπειρογνώμων για το συγκεκριμένο θέμα. Και θέλω να καλωσορίσω επίσης τον Τζουζέπε Νίστικο, ο οποίος είναι εκπρόσωπός μας στον Οργανισμό Φαρμάκων. Κύριε Λούντιν, έχετε ακούσει τη συζήτηση που κάναμε με την κυρία Επίτροπο. Υπήρξαν ορισμένα ερωτήματα τα οποία ουσιαστικά απευθυνόταν σε εσά ως εμπειρογνώμονα. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε τη δική σας άποψη σε σχέση με τα εμβόλια και περιμένουμε αντιμόνως να ακούσουμε τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, έντιμα μέλη. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να προβούμε σε αυτή την ετήσια ανταλλαγή απόψεων. Είναι για μένα η πρώτη φορά που εμφανίζομαι ενώπιον της νέας Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και φυσικά προσβλέπω στο να διατηρήσω την επικοδομητική σχέση που είχα με την προηγούμενη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, είναι μια ευκαιρία η αιτήσια αυτή η ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τα επιτεύγματα του φορέα μας τον τελευταίο χρόνο και να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιον μας. Φυσικά, εφέτος όλη η αιστεία είναι στην πανδημία γρήπης. Είναι ένα θέμα που θα εξακολουθήσει να είναι στο κέντρο της προσοχής των πολιτικών, των μέσων ενημέρωσης και της κοινή γνώμη για τους επόμενους μήνες. Η πανδημία αυτή είναι κάτι για το οποίο υπάρχει προετοιμασία από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Φορέα Φαρμάκου και του Οργανισμού για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών και των άλλων υπηρεσιών της Κομισιόν και των Εθνικών Αρχών εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει αυτές τις προετοιμασίες το 2003, καταρτίζοντας κατευθυντές γραμμές για την φαρμακοβιομηχανία σε σχέση με την ανάπτυξη εμβολίων για πανδημίες γρήπης, με στόχο να εξασφαλίσουμε μια ταχεία εξέταση και έγκριση των ε, εμβολίων από τη στιγμή που ξεκινάει μια πανδημία. Η προκλήση ήταν να μπορέσουμε να έχουμε μια επιστημονική διαδικασία εξέταση η οποία ήταν και ταχεία και ανθεκτικού χαρακτήρα. Ο στόχος, το, η απάντησή μας ήταν λεγόμενη ε, έννοια mock-up, δηλαδή το να έχουμε αρχέτυπα εμβόλια τα οποία επιτρέπουν ένα μεγάλο μέρος του επιστημονικού έργου να γίνουν πριν από την εκδήλωση μιας πανδημίας. Ένα τέτοιο ε, πρωτόλιο, εν πάση περιπτώσει, ή αρχέτυπο εμβόλιο δεν είναι ο στόχος να χρησιμοποιηθεί σε μια πανδημία, παρά μόνο να βοηθήσει να εντοπίσουμε το στέλεχος και να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε τον έλεγχο, ε, το εμβόλιο. Οι μελέτε οι οποίε έχουν γίνει είναι για να εξασφαλίσουν επίση ότι είναι αυστηρέ οι προδιαγραφέ και τα πρωτόκολλα των φαρμακευτικών εταιριών για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ε, εμβολίων και ότι μπορούν να ξεκινήσουν τη δημιουργία αντισωμάτων κατά του ιού. Οι μελέτε οι οποίε έχουν λάβει η χώρα μέχρι στιγμή έχουν περιλάβει 8.000 άτομα μεταξύ των οποίων και ενήλικε και ηλικιωμένα άτομα και παιδιά. Ένα τέτοιο λοιπόν αρχέτυπο εμβόλιο έχει σαν στόχο να προσωμιάσει το τελικό εμβόλιο με δύο τρόπους. Καταρχήν σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή του και για όσο αφορά τη μέθοδο παρασκευής του και σε ό,τι αφορά την λεπτομερή του σύνθεση. Επίσης χρησιμοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ήδη κάποια προστασία εναντίον ενός εναντίον ιού. Από τη στιγμή που έχουμε εντοπίσει το στέρεχος της πανδημίας, μπορούν η παραγωγή των εμβολίων να εισαγάγουν το στέλεχος αυτό στο εμβόλιο και να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ταχεία έγκριση. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται κάθε χρόνο για την έγκριση εμβολίων κατά της ε, εποχικής ε, γρήπης και έχουμε λοιπόν δεκαετίες εμπειρίες με αυτά τα εμβόλια. Έχουμε τέσσερα εμβόλια τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιώντας αυτή τη διαδικασία από το 2007. Ο φορέας μας έχει συν συνιστήσει την έγκριση αλλαγή θελέχους για δύο από αυτά τα εμβόλια την προηγούμενη εβδομάδα στην συνεδρία της Επιστημονικής Επιτροπής 24 Σεπτεμβρίου. Το Φωσέτρια της Νοβάρτης και το Παντεμρίξ της Γκλάξο Σμιθ Κλάιν. Τα εμβόλια αυτά τα οποία ακολουθούν αυτή την προσέγγιση συνιστά τη χρήση τους σε ενήλικα άτομα, μεταξύ των οποίων και τις εγγύους γυναίκες και σε παιδιά από την ηλικία των 6 μηνών. Χρησιμοποιούμε, ε, εργαζόμαστε ακόμα με την Baxter για ένα ακόμα εμβόλιο αυτού του είδους και έχουμε προετοιμάσει μια θετική γνωμοδότηση για τα εμβόλια της ε, Baxter και θα έχουμε τη γραπτή διαδικασία αύριο μαζί με την Επιστημονική Επιτροπή. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα είμαστε σε θέση να λάβουμε μια απόφαση την Παρασκευή, μια θετική απόφαση η οποία μπορεί να διαβιβαστεί λοιπόν στην Κομισιόν, όπως έχει γίνει και η ταχεία διαδικασία έγκρισης για τα δύο προηγούμενα εμβόλια τα οποία ανέφερα. Και μπορεί λοιπόν και το εμβόλιο της Μπάξτερ να έχει την ίδια τύχη την επόμενη εβδομάδα. Η επιτυχία αυτής της διαδικασίας είναι σαφής απόδειξη της ικανότητας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Φαρμάκων να μπορέσει να παράσχει ε, αποτελέσματα σε στενή συνεργασία με την Κομισιόν και τις Εθνικές Αρχές. Η διαφάνεια και η παροχή πληροφοριών είναι ένα βασικό στοιχείο του έργου του φορέα μας. Έχουμε δημιουργήσει μία μικρή ιστοσελίδα μέσα στα πλαίσια της γενικής μας, ε, του δικτυακού μας τόπου, όπου το κοινό και οι υγειονομικοί ε, φορείς μπορούν να βρουν πληροφορίες σε όλες τις γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης εξηγούμε τη διαδικασία αξιολόγησης και τα στοιχεία, τα επιστημονικά, του τη βάση των οποίων γίνονται οι συστάσεις του φορέα μας. Και φυσικά όταν έχουμε νέες πληροφορίες ενημερώνεται αυτή η ιστοσελίδα. Όπως και με όλα τα άλλα φάρμακα είναι απαραίτητο να έχουμε την παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων πανδημίας γρήπης. Από τη στιγμή που αρχίζεται, αρχίζει η χρησιμοποίηση αυτών των εμβολίων, οι παραγωγοί ξεκινούν μία σειρά από πρόσθετες μελέτες που έχουν δεσμευτεί να κάνουν που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια των εμβολίων παρακολουθούν 9.000 άτομα που έχουν νεωστεί εμβολιαστεί για να εξασφαλίσουμε ότι είναι ασφαλή τα εμβόλια ή τα ένα μη ένα. Επίσης, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε και την ανιχνευσιμότητα ώστε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε παρενέργεια μπορεί να ανιχνευτεί στο συγκεκριμένο εμβόλιο και το συγκεκριμένο άτομο το οποίο εμβολιάστηκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση οι φαρμακευτικές εταιρείε που παράγουν αυτά τα εμβόλια θα συνεργάζονται με τις αρχές δημόσιας υγείας για να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα. Το ευρωπαϊκό μας σύστημα έχει ανταποκριθεί στην πρόκληση έγκριση των εμβολίων για την πανδημία. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε όμως ότι οι αποφάσεις για το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα εμβόλια και επίσης η ταυτοποίηση των ομάδων κινδύνου και οι εθνικές εκστρατείε ε, εμβολιασμού είναι αρμοδιότητα των εθνικών αρχών δημόσια υγεία και όχι με τον φορέα φαρμάκων υπηρετικών μισθών. Εμεί εξακολουθούμε να δούμε κατευθυντέ γραμμέ, αλλά η τελική απόφαση για τον εμβολιασμό και το χρονοδιάγραμμά του είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να αντιμετωπίσω άλλο ένα θέμα το οποίο έχει προσελκύσει την προσοχή τη Επιτροπή σα όταν μίλησε το Δεκέμβριο 2008, που είναι το θέμα των αντιβιωτικών και τη αντίσταση στα αντιβιωτικά. Ο φορέα των φαρμάκων και ο Ευρωπαϊκό Φορέα για την Πρόληψη και τον Ελέγχο των Ασθενειών παρουσίασαν τα αποτελέσματα το Σεπτέμβριο του 2009 εργασίας πάνω από δύο ετών που ε, εξέτασε το χάσμα μεταξύ των μολύνσεων που προέρχονται από βακτηρίδια τα οποία είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά και τη ανάπτυξη νέων αντιβιωτικών που θα τα αντιμετωπίσουμε. Τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα μα. Ούτε είναι ενθαρρυντικά τα πορίσματα, ούτε όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε. Το πόρισμα της έκθεσης είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ του, των, <clears throat> του αριθμού των μολύσεων που προέρχονται από πολλαπλά ανθεκτικά βακτηρίδια και της ανάπτυξης νέας γενιάς αντιβιωτικών. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πορίσματα είναι ότι περίπου 25.000 ασθενείς πεθαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μολύνσεις με συγκεκριμένα βακτηρίδια που είναι ανθεκτικά, που είναι πολλαπλώς ανθεκτικά και αυτή η αντίσταση αυξάνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μεταξύ των βακτηριδιών που είναι γκραμ αρνητικά. Η έκθεση θεωρεί ότι οι μολύνσεις από αυτά τα πολλαπλά ανθεκτικά βακτηρίδια οδηγούν σε πρόσθετο άγχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, μαζί με την απώλεια παραγωγικότητα. Τα αποτελέσματα αυτή τη μελέτη παρουσιάστηκαν σε μια ειδική διάσκεψη που οργάνωσε η Σουηδική Προεδρία στι 17 Σεπτεμβρίου 2009 και έχουν επίση διαβιβαστεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια στρατηγική και επίση και μια παγκόσμια στρατηγική να αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσει αυτό το χάσμα. Ο Ευρωπαϊκό Φορέα ε, Φαρμάκων και η ECDC είναι έτοιμε να παίξουν το ρόλο του για την εφαρμογή αυτή τη στρατηγική, η όθηση για την οποία όμω θα πρέπει να έρθει από τι πολιτικέ αρχέ. Και ξέρω ότι η Σουηδική Προεδρία έχει ήδη θέσει μια προτεραιότητα σε αυτό το επίπεδο. Ελπίζω λοιπόν ότι η Σουηδική Προεδρία θα προωθήσει το θέμα αυτό και κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Υγεία τον Οκτώβριο. Επομένω, νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ, διότι και θα υπάρχουν πολλές ερωτήσεις και κύριε Πρόεδρε, Έχω ήδη ακούσει ορισμένα από τα ερωτήματα. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να απαντώ, να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα ή αν θα πρέπει να περιμένω και τις περαιτέρω ερωτήσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κύριε Λούντριεν για τις πληροφορίες σας. Νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε στους συναδέλφους που θα θέσουν ερωτήματα και ίσως εσείς μπορείτε να προσθέσετε και στοιχεία τα οποία δεν περιέχονται σε αυτές τις ερωτήσεις, αν το θεωρείτε αυτό σκόπιμο. Κύριε Κροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί τα έχουμε πει τα περισσότερα. Το Βασικό είναι να έχουμε σωστές πληροφορίες από τις κατάλληλες πηγές. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή που ήρθε σήμερα εδώ. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε μια επιταχυμένη διαδικασία για την έγκριση αυτών των εμβολίων, γιατί έχουμε χάσει πολύ χρόνο όμως θα έπρεπε αυτή η διαδικασία να χρησιμοποιείται για τα γενικά φάρμακα. Γιατί όταν έχουμε ένα νέο φάρμακο που πρόκειται να εγκριθεί για διάθεση στην αγορά και το οποίο είναι νέο φάρμακο, πάλι θα έπρεπε να το έχουμε στη διάθεσή μας το συντομότερο δυνατόν. Αυτό ως ξεχωριστή σκέψη μου. Τώρα, όσον αφορά τις δόσεις, που προβλέπονται για τον εμβολιασμό. Εσείς προτείνετε έναν εμβολιασμό. Όμως στο παρελθόν στη χώρα μου είχαν σκεφτεί ότι θα έπρεπε να παραγγείλουμε δύο δόσεις ανά κάτοικο οι οποίες θα έπρεπε να γίνονται με κάποιες ημέρες διαφορά. Θα ήθελα λοιπόν κάποιες διευκρινήσεις εδώ. Και τέλος ένα ερώτημα που πιστεύω ότι απασχολεί και άλλους συναδέλφους. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιες πληροφορίες για τα adjuvants, τα βελτιωτικά, τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται. Θεωρείτε ότι όντως είναι μηδενικός ο κίνδυνος. και ότι το εμβόλιο είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιουσδήποτε κινδύνους μπορεί να προκύψουν από αυτά τα βελτιωτικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά. Ευχαριστούμε κυρία Γκροστέτ ή κυρία Ροτμπέραντ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε η κυρία Γκροστέτ ε, και μετά από αυτά που είχαν ήδη ρωτήσει κάποιοι συνάδελφοι την κυρία Βασιλείου παρόλο που δεν είναι δική της αρμοδιότητα θα ήθελα να επανέλθω στη διαδικασία πρέπει να τονίσουμε ότι η διαδικασία για τα φάρμακα έχει μία νομική βάση, έχει αποφασίσει επ' ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι κάτι που αποφασίζουμε εμείς και όχι οι φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη νομική διαδικασία που έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς δεν θέλουμε να δεχτούμε κινδύνους για την υγεία. Οπότε, όσον αφορά την επιταχυμένη διαδικασία, προκαλεί αντιδράσεις και προκαλεί φόβο. Το ακούσατε και εδώ, το έχετε ακούσει υποθέτω και γενικά. Τι πρέπει να αναμένει από αυτό ο κόσμος. Θα υπάρξουν ωφέλη, θα είναι μεγαλύτερες οι παρενέργειες και πιο ανεξέλεγκτες από ό,τι σε σχέση με άλλα εμβόλια όπως αυτά για την εποχιακή γη πρέπει. Και επίσης πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της εποχικής γρήπης και το εμβόλιο για την H1N1, γιατί δεν πρέπει να λέμε πλέον γρήπη των χείρων, από ό,τι λέει ο συνάδελφος, γιατί μπορεί να υπάρξει πρόβλημα με την κτηνοτροφία. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν το εμβόλιο για το H1N1 γιατί είναι ανεξέλεκτες οι παρενέργειες. Τέλος, όσον αφορά τα αντιβιωτικά, δεν ξέρω τι να πω. Και εγώ και άλλοι συνάδελφοι το επαναφέρουμε αυτό το θέμα τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια. Και πάντα λέμε δεν έχουμε αρκετά προβλήματα με την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά και τα αντιμικροβιακά. Γνωρίζουμε ότι αυξάνεται η ανθεκτικότητα δεν ήξερα τα ακριβή νούμερα, 25.000 λέτε, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί θάνατοι εξαιτίας της ανθεκτικότητας στα βακτήρια. Και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και νοσοκομεία που βρίσκονται σε μαύρη λίστα που θα έπρεπε να κλείσουν. Παρόλα αυτά υπάρχουν αυτές οι μαύρες λίστες όπου μπορούν να μάθουν οι ασθενείς τι αριθμός βακτηρίων υπάρχει σε ένα νοσοκομείο. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Οπότε, αυτή τη στιγμή τα αντιβιωτικά, τα οποία δεν τα παράγουμε εμείς ως κοινοβούλιο, ούτε η ΕΜΕΑ, τα παράγουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Και πραγματικά δεν θεωρώ ότι χρειάζονται κίνητρα για την παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Χαίρομαι που τονίσατε την σημασία της Σουηδικής Προεδρίας, αλλά πρέπει να αποφασίσουν τι θα γίνει με τα αντιβιωτικά. Θα κάνουμε φοροαπαλλαγές στα κράτη-μέλη, θα έχουμε επιταχυμένη διαδικασία έγκρισης. Πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Γνωρίζουμε ότι κάποια αντιβιωτικά δεν θα είναι τόσο αποδοτικά οικονομικά. Τι θα κάνουμε για να δώσουμε κίνητρα στις βιομηχανίες. Σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις καλές ερωτήσεις σας. Κυρία Πιλάρα Γιούσο έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ πολύ σύντομη σε σχέση με την ερώτηση της κυρίας Ροντ Μπέρετ για την ασφάλεια του εμβολίου. και για τότε θα έχουμε παρενέργειες. Ξέρετε ότι μέρος του υγειονομικού προσωπικού αρνείται να εμβολιαστεί. Γιατί πολλοί θυμούνται της παρενέργειας ε, του εμβολίου με το στέλεχος της κλινικής Μάγιο ε, στο παρελθόν. Ε, πάλι πρόκειτο για ένα στέλεχος της γρήπης των χείρων. Και αυτό, και αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο περιέχει τέτοια στελέχη. Γι' αυτό ανησυχούν πολύ. Γιατί θυμούνται αυτό αυτές τις παρενέργειες που προήλθαν από αυτό το εμβόλιο τότε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Μπορείτε να μας ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα νευρολογικής φύσεω, καμία παρενέργεια. Και επίση να σα ρωτήσω την άποψή σα για τον εμβολιασμό παιδιών κάτω των 14 ετών. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων στου παιδιάτρους. Merci. Vous avez Ωραία. Τελειώσατε, ναι. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά που είσαστε μεταξύ μας. Εγώ πήγα και έψαξα στο δικτυακό σας τόπο στο ίντερνετ και ψάχνω πάντα να βρω για αυτές τις περίφημες βελτιωτικές ή ενισχυτικές ουσίες, τα adjuvant. Εγώ δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει κάτι εκεί. Τα έκτοχα. Αναφέρεται λοιπόν διάφορε ουσίε όπω είναι το τσουμεσόλ, το οποίο έχει, περιέχει υδράριο, και δεν λέτε τίποτα για τα έκδοχα. Εγώ απευθύνθηκα λοιπόν κατευθείαν στην Νόβαρτης που μου λέει ότι χρησιμοποιούν σκουαλέν γιατί ξέρουν ότι το αλουμίνιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρενέργειες και χρησιμοποίησαν αυτό το εμβόλιο για να χρησιμοποιήσουν ε, ένα, ε, να χρησιμοποιήσουν μια ουσία που προέρχεται από, από λίπος ε, καρχαρία. Την έχουν βάψει οι καρχαρίες λοιπόν, λέω παρενθετικά. Αλλά ποιε είναι οι παρενέργειε που μπορεί να προέρχονται από, από αυτήν την ουσία. Στον πόλεμο του Περσικού κόλπου υπήρχε τότε πάλι ένα εμβόλιο που είχε την ίδια αυτή ουσία που προέρχεται από το λίπο των καρχαριών. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια σύνδεση για τα δύο. Επίση για τον Μπάξτερ. Εγώ είδα την αγωγή η οποία έχει γίνει από μία δημοσιογράφο σε σχέση με αυτό το εμβόλιο που κατετέθη πέρσι. Εσείς έχετε παρέμβει σε επίπεδο της ΕΜΕΑ, του Οργανισμού Φαρμάκων για αυτό το φάρμακο. Ήταν μια Αυστριακή δημοσιογράφος που εστράφη κατά της Μπακτέρ και της Αβίρ Ιλ. Αυτό ήταν ένα φάρμακο το οποίο είχε διανεμηθεί στην τσεχική δημοκρατία. Τι μπορείτε να μας πείτε σε σχέση με αυτήν την υπόθεση. Τρίτον, για το ερωτηματολόγιο χρήσης που θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν οι ιατροί και οι νοσοκόμες εμβολιάσουν παιδιά κτλ. Έχετε προβλέψει σε αυτό το ερωτηματολόγιο να τίθενται ερωτήματα σε σχέση με, την, με το αν είναι αλλεργικά για τις πρωτεΐνες των πουλερικών τα παιδιά. Γιατί αυτό το εμβόλιο έχει καλλιεργηθεί σε υπόβαθρο από πρωτεΐνες πουλερικών. Και τέλος, για τη στρατηγική που ακολουθείτε. 24 Απριλίου 2009 εμφανίστηκε αυτό το, <clears throat> αυτή η ασθένεια. Όταν λέτε αρχή πρόληψης, να αποφύγουμε την πανδημία, όταν λέτε μπορεί να φτάσει στο 30% το ποσοστό του πληθυσμού που θα μολυνθεί. Το καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια σωστή αντιμετώπιση σε επίπεδο στρατηγικό. Τώρα όμως έχουμε τις πληροφορίες για το τι έγινε στην Αυστραλία και στην Αργεντινή. Στην Αυστραλία 20 εκατομμύρια άτομα είναι ο πληθυσμός μόνο 5% έχει μολυνθεί και κάποιες εκατοντάδες νεκρών. Ίσως δεν έπρεπε να πεθάνω αυτοί, το καταλαβαίνω, αλλά σε σχέση με την εποχική γρήπη είναι πολύ μικρό ποσοστό. Στην Αργεντινή 40% πληθυσμό 2,5% του πληθυσμού μολύνθηκε, 400 με 500 θάνατοι, καμία σχέση και πάλι σε σχέση με αυτούς που, θανάτους που προέρχονται από την εποχική γρήπη. Με την απόσταση λοιπόν τη χρονική που έχουμε τώρα πια μήπως θα έπρεπε να επανέλθουμε σε μια πιο λογική αντιμετώπιση λέγοντας ούτως ή άλλως ο ιός αυτός βρίσκεται στην Ευρώπη, στη Γαλλία, η Γαλλία ίσως είναι η πιο μολυσμένη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, υπάρχει αυτός ο ιός, είναι μια πλήρως ανώδυνη γρήπη, δεν υπάρχει λοιπόν λόγος πανικού και μαζικού εμβολιασμού αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση για μια μαζική μορφή εμβολιασμού, αλλά για αυτούς που έχουν καρδιοαγγειακά προβλήματα, προβλήματα νεφρικά, αναπνευστικά ή παχυσαρκία, ίσως εκεί έχει νόημα να <clears throat> εμβολιαστούν τα άτομα αυτά. Σήμερα το εμβόλιο για την εποχιακή γρήπη δεν έχει έκδοχα, ενώ το εμβόλιο για την ΙΤΑ 1 έχει έκδοχα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα εμβόλια. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε Κύριε Λαντρίν, θέλετε να πείτε κάτι σε σχέση με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Σας ε, ευχαριστώ. Πρέπει να όλα μια προοπτική χρονική σε όλα αυτά. Η πανδημία αυτή ξεκίνησε τον Απρίλιο αυτού του έτους. Δεν έχουν περάσει και πολλοί μήνες από τότε. Το στέλεχος εντοπίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που δήλω, ε, ε, κήρυξε την επιδημία το Μάιο νομίζω. Και τον Ιούνιο είχαμε το στέλεχος και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να παράγουμε το, το στέλεχος. Πήγαμε, απευθύνθηκαμε σε όλα τα εργαστήρια, φαρμακοβιομηχανίες Είναι προφανές ότι δεν έχουμε κλινικά δεδομένα γιατί πρόσφατα ανακαλύφθηκε αυτό το στέλεχος. Αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν έχουμε κλινικά δεδομένα για τα εμβόλια που έχουμε σήμερα. Ήμασταν τυχεροί στην Ευρώπη γιατί ακολουθήσαμε αυτή την, ε, την τακτική mock-up. Ε, έχουμε λοιπόν ένα εμβόλιο που, που παρήχθη με τις καλύτερες, με τις βέλτιστες φαρμακευτικές ε, διαδικασίες παραγωγής, με παρόμοιο στέλεχο με τη γρήπη των πτηνών και βεβαίως χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να προβάλλουμε τη, γνώση αυτών κλινικο, από αυτές τις κλινικέ δοκιμές του παρελθόντο σε αυτό το νέο στέλεχο, σε αυτό το νέο εμβόλιο. Αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο με την εποχική γρήπη. Δεν είναι τελείω καινούριο εμβόλιο. Είναι σαν το εμβόλιο της εποχικής γρήπη, αλλά με ένα νέο στέλεχος ε, για το οποίο το μεγαλύτερο μέρος ε, του πληθυσμού ε, δεν έχει ανοσία. Δεν έχουμε λοιπόν κλινικά δεδομένα για αυτό το συγκεκριμένο στέλεχος. Τώρα, μπορείτε να κάνετε ένα υπολογισμό για τον κίνδυνο που αναλαμβάνουμε. Εάν καθυστερήσουμε την εμπορία του εμβολίου αυτού, θα μπορούσα να σας πω ότι αν κάνετε αυτόν τον υπολογισμό, θα δείτε ότι η πλάστικα σαφώς θα γέρνει υπέρ του να τεθεί στην αγορά και να αρχίσει ο εμβολιασμό. Σε σχέση με μια άλλη κατάσταση όπου θα περιμέναμε για να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Ο κίνδυνος για παρενέργειες από αυτό το εμβόλιο είναι ελάχιστο σε σύγκριση με αυτούς που θα μολυνθούν από τον ιό στο μεταξύ χρονικό διάστημα και που ενδεχομένως πεθάνουν από την πανδημία. Άρα, αυτή είναι η ερμηνεία που δίδουν όλες οι υγειονομικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων και των υπόλοιπων υγειονομικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να ζυγίσουμε τα πλεονεκτήματα, τα ωφέλη και το, την πιθανότητα την πολύ μικρή πιθανότητα παρενεργειών, ανεπιθύμητων ενεργειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα, η Ντάγμα Ροντμπέρετ μίλησε για τη διαδικασία για την άδεια εμπορία. Συμφωνώ για την έγκριση εμπορία. Πρέπει να είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία για τις εγκρίσεις και για την επιστημονική αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα διαβεβαιώ, δεν μα τα υπαγορεύουν όλα αυτά. Δεν είμαστε οι φαρμακοβιομηχανίε. 20% ε, από τι αιτήσει τι απορρίπτουμε. Η διαδικασία μας είναι ε, απόλυτα αδιαπερατή. Τώρα, έγιναν ορισμένε ερωτήσει που αφορούν τη δόση. Μία δόση ή δύο. Οι συστάσει προ στιγμή, με βάση την εμπειρία που είχαμε με δοσολογία του πειραματικού εμβολίου του ΜΟΚΑΠ και την προβολή ε, και, ε, καταλήξαμε λοιπόν από τις κλινικές δοκιμές με το εμβόλιο ΜΟΚΑΠ στο ότι απαιτούνται δύο δόσεις. Καταλαβαίνετε βεβαίως ε, ότι συνεχίζουν οι κλινικές δοκιμές και περιμένουμε κάθε μέρα τα αποτελέσματα αυτών των κλινικών δοκιμών. Μόλις θα έχουμε πιο αξιόπιστα στοιχεία για τη δόση, η Επιτροπή θα επαναξετάσει το ζήτημα του κατά πόσο απαιτείται μία δόση ή δύο δόσεις και θα, ενδεχομένως ε, θα κάνουμε νέες συστάσεις. Τώρα για αυτά τα adjuvants, τα βελτιωτικά, τα ενισχυτικά. Υπάρχει μεγάλη εμπειρία για τη χρήση τους. Και είναι πολλά τα ωφέλη. Πρώτα απ' όλα, μειώνεται ε, η ποσότητα του του, του ιού ε, κατά τέσσερις φορές λιγότερο ε, του ιού που τύφεται στο εμβόλιο. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ σημαντικό σε περίπτωση πανδημίας, όπου είναι σημαντικό όσο να τον πιο γρήγορα να βρούμε αρκετό ιό για να ξεκινήσουμε το εμβολιασμό. Αν θέλουμε τετραπλάσια δόση, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τόσα πολλά εμβόλια. Επίσης, τα ενισχυτικά αυτά ε, προκαλούν πολύ καλύτερη ανοσοαπόκριση. Άρα υπάρχουν θετικές πτυχές, ε, πολλά τα ωφέλη, γι' αυτό χρησιμοποιούνται ευρέω. Όχι μόνο στο εμβόλιο της γρήπης, αλλά και σε άλλα εμβόλια. Τώρα, αυτά τα, τα στοιχεία δεν είναι επικίνδυνα χημικά. Το σκουραλένιο, για παράδειγμα, είναι μια φυσική ουσία που την έχει ο οργανισμό μας. Ε, στις κυταρικές μεβράνες των κυτάρων. Είναι φυσική ε, ουσία που βρίσκεται στα κύτταρά μας. Ε, και σε ένα εμβόλιο GSK DSKV ε, που είναι ε, βιταμίνη K. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα ε, με τη χρήση τους. Έγινε μία ερώτηση για την ασφάλεια σε σχέση με αυτά που έγιναν το 76 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω ότι αυτό ήταν τελείως διαφορετικό εμβόλιο. και ποτέ δεν αποδείχθηκε ότι υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα σε αυτές τις νευρολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες και στο εμβόλιο. Ήταν, ήταν βεβαίως τέλεχος ε, νη ένα ή τα 1 και τέτοια στελέχη συμπεριλήφθηκαν και στο εποχιακό εμβόλιο για πολλά χρόνια. Το εμβόλιο της εποχιακής γρήπης. Και ποτέ δεν παρουσιάστηκαν τα φαινόμενα που παρουσιάστηκαν το 1976 στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και το εξετάσαμε αυτό, εξετάσαμε τα ωφέλη από το εμβόλιο. Παρ' όλα αυτά, σα το λέω και είναι σημαντικό. Θέλουμε ένα αξιόπιστο σύστημα follow-up για να δούμε αν υπάρξουν ιδιαίτερα παράξενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αν υπάρχουν, ακόμα και αν υπάρχουν, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τι ανακαλύψουμε άμα δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμός γιατί θα είναι τόσο μικρή ε, η συχνότητα εμφάνισης των ε, παρενεργειών που θέλουμε μεγάλη έκθεση, έκθεση μεγάλου μέρους του πληθυσμού για να μπορέσουμε να τα δούμε. Να δούμε τις παρενέργειες. Δεν, δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν παρενέργειες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα πολύ αξιόπιστο σύστημα follow-up και με ανεξάρτητε μελέτες και με μελέτε που διεξάγονται από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και να σας πω και το εξή. Αυτές οι μελετες follow follow-up για τη χρήση των εμβολίων ε, και, και, και σε σχέση με την κλινική πραγματικότητα δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στενότητα συνεργασία και με τον υπόλοιπο κόσμο και με τι Αμερικανικέ αρχέ και με άλλε αρχέ στον υπόλοιπο κόσμο. Με τι αρχέ τη Αυστραλία που προφανώ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χειμώνα του και άρα συνεχίζεται η επιδημία εκεί. Λοιπόν, απάντησα για τη δόση. Μίλησα και λίγο για τα για αυτά τα ενισχυτικά. Σα είπα για το τι έγινε το 76 στι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε το θέμα των ελληνικών εντράσεων. Ναι, ε, στο, στις πληροφορίες για το προϊόν αναφέρεται μέσα στο έντυπο ότι αυτοί που είναι ε, αλλεργικοί ε, σε πρωτεΐνη αυγού, δεν, σε αυτούς αντενδείκνυται το εμβόλιο. Είναι θέμα λοιπόν και των εμβολιαζομένων, ε, αλλά κυρίω των, των ιατρών που θα εμβολιάσουν, του υγειονομικού προσωπικού που πρέπει να ρωτήσουν το άτομο το οποίο θα κάνει το εμβόλιο, είναι αλλεργικό στην πρωτενη αυγού. Αυτό αναφέρεται και στι προδιαγραφέ και στι οδηγίε για το προϊόν. Α, ε, όσον αφορά την Baxter, είχε αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, τα εξετάσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και βεβαίως ελήφθησαν υπόψη. Αυτή την εβδομάδα είχαμε εξωτερικό έλεγχο στι εγκαταστάσει τη Baxter για να είμαστε 100% σίγουροι ότι η παραγωγή ε, θα είναι 100% αυτή που θα έπρεπε. Ε, ήταν άκρο θετικά αυτή τα αποτελέσματα, γι' αυτό και περιμένουμε να είναι θετική γνωμοδότηση για την Baxter. Τέλος, η Dagmar μου είπε να αναφερθώ στο θέμα της, ε, της, ε, ε, των αντιβιωτικών και τη αντίσταση στα αντιβιωτικά. Μα κοιτάξτε, αν η, επιχείρη, αν η, φαρμακοβιομηχανία δαπανά 100 δολάρια στην έρευνα για το αντιβιωτικό, θα 100 δολάρια θα πάρει πίσω. Και αν αποφασίσει να επενδύσει κάπου αλλού, θα τα επενδύσει κάπου αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι. Ε, αναπτύσσουν ε, ε, από τη μια. Ε, αν, αν παρασκευάσουν αντιβιωτικά, δεν θέλουμε να τα ρίξουμε στο εμπόριο, γιατί δεν θέλουμε να, τα, να παίρνουμε και στα μαζικά και να υπάρξει αντίσταση και σε αυτά. Άρα, καταλαβαίνετε, δεν, δεν περιμένουν να διατεθεί σε ευρέω στην αγορά το καινούριο αντιβιωτικό ταυτόχρονα ε, μην ξεχνάμε, θα κοστίσει ιδιαίτερα η παραγωγή νέων αντιβιωτικών. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κάποια κίνητρα στις φαρμακοβιομηχανίες για να αναπτύξουν νέες, ε, νέου είδους ε, αντιβιωτικά. Και αυτό σίγουρα ε, συζητήθηκε και στη συνεδρίαση της ειδική Προεδρίας και στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, Σουηδία. Και από ό,τι ξέρω, μάλλον θα κάνει κάποια συγκεκριμένη πρόταση η Σουηδία για το πώ θα λυθεί το πρόβλημα. Τώρα, εγώ έχω κάποιε ιδέε στο μυαλό μου αλλά επειδή εμεί δεν χαράσουμε πολιτική ω οργανισμό για τα φάρμακα, δεν πρόκειται να χώσω τη μύτη μου σε αυτή την υπόθεση. Ευχαριστώ, ο κύριος Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Λούντγκεν. Εμείς τώρα έχουμε, όπως είπατε, αντενδείξεις σε περίπτωση αλλεργίας στο λεύκομα Υπάρχουν άλλες ε, αντενδείξεις, υπάρχουν άλλες ομάδες πληθυσμού όπου εσείς θα, προ... θα συνιστούσατε να μην γίνει κάποια... κάποιος εμβολιασμός και υπάρχουν κάποιες... Ε, κάποιοι περιορισμοί για, τα... για τον εμβολιασμό. Υπήρξε το ερώτημα αυτό για τις εγγύους στο πρώτο τρίμηνο. Υπάρχει κάποιος περιορισμός της έγκρισης. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε σαφείς. Γιατί ήδη αν εμείς είμαστε μπερδεμένοι μετά από αυτά που ακούσαμε την κυρία Γιάκαμπ, όπου αναφέρθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα για τα παιδιά και για τις ομάδες, κάποιες ομάδες κινδύνου. Φανταστείτε πόσο μπερδεμένοι πρέπει να νιώθουν οι απλοί άνθρωποι. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν η έγκριση αυτών των δύο εμβολίων περιλαμβάνει περιορισμούς για ορισμένες ομάδες πληθυσμού για τις οποίες δεν ισχύει η έγκριση αν Υπάρχει λοιπόν <clears throat> μια έγκριση για ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά ή οι έγκυες και ένα δεύτερο σημείο το θέμα των, ε, της αντιμετώπισης με πολυϊκά φάρμακα όπως είναι το ταμιφλού. Είναι δυνατόν να ανοίξει ένα παιδί την κάψουλα και να την περιεργαστεί. Ε, στη δική μου κλινική εμπειρία θα πρέπει οι γονείς να αναλαμβάνουν την ευθύνη να ανοίγουν την κάψουλα και να δίνουν τα, το περιεχόμενό της στα παιδιά. Δεν ξέρω λοιπόν αν η, ο μέσος γονέας ξέρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η παροχή αυτού του σκευάσματος προς το παιδί. Μπορεί κάποιος γονέας να μην ξέρει καλά τη γλώσσα στην οποία ζει, να μην μπορεί να διαβάσει λοιπόν τις οδηγίες. Εγώ έχω πολλές αμφιβολίες για το αν είναι αυτή η σωστή αντιμετώπιση των παιδιών και θα ήθελα να έχουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο παροχής αυτού των φαρμακών προς τα παιδιά. Ευχαριστώ κύριε Λίζε. Η κυρία Μακίβαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο ερώτημα για τα ενισχυτικά, τα που δεν συνδέεται άμεσα με το θέμα της ε, γρήπης, αλλά το οποίο έχει αναφερθεί στα μέσα ενημέρωση στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη βδομάδα ένα νεαρό κορίτσι πέθανε μερικές ώρες μονάχα αφού της κάνανε το εμβόλιο για τον, τράχυλο της, για τον καρκίνο του τραχύλου της ε, μήτρας. Ήταν 14 χρονών. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ του εμβολίου και του θανάτου της. Είπα ο γιατρός ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ήταν το σεβαρίξ το φάρμακο αυτό. Ορισμένοι είπανε ότι το... η ενισχυτική ουσία που χρησιμοποιείται στο Σεβαρίξ είναι η ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στο εμβόλιο για τη γρήπη H1N1. Μπορείτε να το διευκρινίσετε αυτό. Euh, Με συγχωρείτε. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να σηκώνει το χέρι του, άρα αυτό ήταν το τελευταίο ερώτημα. Παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις και να συνοψίσετε. Ευχαριστώ. Όσον αφορά το Σεβαρίξ, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι δεν πρόκειται για την ίδια ενισχυτική ουσία. Ωστόσο, σημειώσαμε αυτή την περίπτωση. Θα υπάρξει έκθεση παρενεργειών που θα σταλεί στην ΕΜΕΑ για αυτό το θέμα του Σεβαρίξ. Πάντως, μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από εκατομμύριο δόσεων που έχουν χορηγηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα πρέπει να τα υπόψη μας και αυτά. Από την άλλη πλευρά όμως συνεχίζεται το έργο μας για να κατανοήσουμε την υπόθεση. Τώρα όσον αφορά το ταμιφλού. Όντως η κατάσταση είναι δύσκολη όσον αφορά τα παιδιά. Πάντως συζητήσαμε το θέμα στην Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη στιγμή επεκτείνουμε την ενδείξεις για το ταμιφλού για παιδιά μικρότερα από τους 6 μήνες σε περίπτωση πανδημιών. Άρα μειώσαμε το όριο ηλικίας. Βεβαίως είναι δύσκολο το θέμα γιατί δεν έχουμε παιδιατρική εκτίμηση. Παρόλα αυτά αυτό που κάναμε είναι να να καταλήξουμε σε ειδικά σκευάσματα για τα παιδιά μικρότερα του ενός έτους. Όμως, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σκευάσματα ειδικά παιδιατρικά, θα υπάρξει πρόβλημα συμμόρφωσης. Ίσως θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των φαρμακοποιών για την παρασκευή αυτών των σκευασμάτων, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να βοηθήσουν οι φαρμακοποιοί τους γονείς. Ίσως λοιπόν πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να καταλήξουμε στη σωστή δοσολογία, στο σωστό σκεύασμα. Και Ίσως θα μπορούσα να δώσω το λόγο στον εμπειρογνώμονά μου, τον κύριο Καβαλιέρη, για να μιλήσει για το θέμα των παιδιών και των εγγύων. Ευχαριστώ, Τόμας. Όσον αφορά τα παιδιά, οι συστάσεις που αναφέρονται στις πληροφορίες προϊόντος βασίζονται ουσιαστικά στο σχέδιο εμβολίου που είχαμε κάνει για το H5N1 και γι' αυτό είχαν γίνει κλινικές μελέτες, οι οποίες κλινικές μελέτες είναι η βάση για τις συστάσεις που κάνουμε για το H1N1. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αντένδειξη και δεν μπορούμε να κάνουμε σύσταση για παιδιά μέχρι έξι μηνών. Δεν μπορούμε να κάνουμε συστάσεις για αυτά γιατί δεν έχουμε εμπειρία ούτε για το εμβόλιο, για την κανονική γρήπη, για αυτή την ηλικία ομάδα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες ηλιακές ομάδες, αυτό που βρήκαμε για τα παιδιά μέχρι 17 ετών είναι ότι είναι δυνατόν να γίνει εμβολιασμός με την κανονική ενόλη ενήλικη δόση. Τα δεδομένα που έχουμε για το H5N1 για την ηλιακή ομάδα 3 έως 9 έτη είναι μισή δόση και άρα η ECDC θεωρεί ότι για την ηλικία 3 έως 9 ετών και για 6 μηνών έως 3 ετών θα προτείνουμε μισή δόση, ενώ για τις ηλικίες 9 έως 17 θα προτείνουμε την ενήλικη δόση. Αυτά γνωρίζουμε προς το παρόν όσον αφορά τα παιδιά. Σε αυτά τα συμπεράσματα έχουμε καταλήξει όσον αφορά τη δοσολογία. Τώρα, όσον αφορά τις ε, εγκύους. γνωρίζουμε από τις ανασολογικές δοκιμές που έχουν γίνει σε εγκύους με το εμβόλιο της κανονικής γρήπης, δεν θεωρούμε ότι θα υπάρξει διαφορά για τις εγγύους. Μπορούμε να κάνουμε λοιπόν κάποιες προβολές. Τώρα βεβαίως όσον αφορά την ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή στις ΙΠΑ πολλές έγκυες κάνουν το εμβόλιο για την κανονική γρήπη. Για παράδειγμα, 2 εκατομμύρια γυναίκες είχαν κάνει το εμβόλιο την περίοδο 2000 έως 2003. Οπότε, με βάση αυτά τα στοιχεία και με βάση κάποιες ε, μελέτες που έχουν γίνει σε ζώα θεωρούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι ασφαλές αυτό το εμβόλιο για τις εγκύους γυναίκες. Παρόλα αυτά ε, βρίσκονται σε εξέλιξη τέτοιου είδους δοκιμές. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν οι απαραίτητες προφυλέξεις και η ΕΜΕΑ έχει έρθει σε επαφή και με την ΕΣΥΝΤΙΣΗ και με τις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου να υπάρξει συνεργασία για παράδειγμα με το δίκτυο για τις ε, γενετικές ε, ανομαλίες προκειμένου να δούμε αν υπάρχει περίπτωση προβλημάτων με αυτό το εμβόλιο. Και, να σας πω ότι έχουμε δώσει, έχουμε δώσει ήδη μια θετική γνωμοδότηση για τρία εμβόλια τύπου mock-up, τρία αρχέτυπα εμβόλια, αλλά τώρα αρχίζει το πραγματικό έργο μας να δούμε τι γίνεται όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα εμβόλια και ο οργανισμός φαρμάκων κάνει ό,τι είναι δυνατό για να έχουμε ένα σύστημα ταχείας αντιμετώπισης οποιασδήποτε παρενέργειας και είμαστε απόλυτα διαφανείς όταν έχουμε πληροφορίες θα τις διαβιβάσουμε και σε εσάς και θα γίνουν βέβαια και οι κλινικές μελέτες στα παιδιά και τις έγκυες στις γυναίκες και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή της δοσολογίας και σε άλλα θέματα. Θα είναι ε, ενήμερο το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Νηστικός ήθελε να παρέμβει. Ε, Που είναι εκπρόσωπός μας ε, στον οργανισμό φάρμακων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ως μέλος της Επιτροπής αυτής είμαι πραγματικά υπερήφανος όταν ακούω τα ειδικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν ευχαριστώ την κυρία Γκροστέ, την κυρία Ροτ Μπέρεντ, τον Πίτερ Λίζε, την Πιλάρ Αϊούζο και επίσης τα ερωτήματα αυτά αντιμετωπίζουν και ειδικά θέματα πολλές φορές αλλά επειδή και εγώ είμαι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής θέλω να ευχαριστήσω αυτούς τους συναδέλφους για το δίκτυο αριστείας το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους εμπειρογνώμονες που δουλεύουν μέρα και νύχτα και πράγματι έχουν την ευθύνη Όπω η Ρίκα Ντίμιν, ο τόμα Άτσεν από την ε, Σουηδία και ορισμένα άλλα άτομα που έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θέλω να τονίσω ότι είναι καθήκον όλων τους θα πρέπει τα μέλη του Κοινοβουλίου να είναι ευτυχή και υπερήφανα που έχουν τέτοια αξιόλογα άτομα στην Επιστημονική Επιτροπή. Και πάντα ακολουθούμε την αρχή της πρόληψης. Για όλα αυτά τα θέματα τα μπορούν τα οποία μπορεί να ανακύψουν για οποιοδήποτε ε, πρόβλημα, οποιαδήποτε παρενέργεια. Πράγματι θα πρέπει να είσαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια στρατηγική και να εξετάσουν τα άτομα τα οποία είναι εκτεθειμένα σε ένα κίνδυνο εκ των υστέρων, εξ και θα πρέπει να αποκομίσουν περισσότερα στοιχεία για το όφελος του γενικού πληθυσμού. Θέλω να πω επίσης όμως ότι πρέπει να αποφύγουμε <clears throat> πανικό και γενική ανησυχία. Γιατί βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τρομοκρατούν τον κόσμο. Βάσει των στοιχείων που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα εμβόλια είναι απόλυτα ασφαλής. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό σε σχέση με το σκουάλεν, το ενισχυτικό αυτό. Το σκουάλεν απλώς μειώνει τη χολυστερίνη. Δεν είναι τοξικό. Είναι, είναι ένα γαλάκτομα. Ελαιόδες γαλάκτομα. Δεν έχει γενετικές ιδιότητες, απλώς ενισχύει τις γενετικές ιδιότητες του εμβολίου. Για το θειομέρσαλ που έχει εθιλικό υδράργυρο. Αυτό πράγματι έχετε δίκιο, θα μπορούσε να είναι δυνητικά επικίνδυνο γιατί είναι μια νευροτοξική ουσία. Αυτό το βαρύ μέταλλο μπορεί να προκαλέσει νευροτοξικά αποτελέσματα, αλλά η δοσολογία η οποία είναι παρούσα στα εμβόλια είναι τόσο μικρή, μόνο 25 μιλιγκράμμ και πιστεύω ότι θα πρέπει να παρακολουθήσετε το θέμα αυτό σε άλλα επίπεδα. Εδώ έχετε μονάχα δύο φορές 25 μικρογραμμάρια διορθώνει ο ομιλητής, ενώ στα τρόφιμα η Επιτροπή Περιβάλλοντος το γνωρίζει καλά, υπάρχει συνεχής παρουσία αυτών των ουσιών στα τρόφιμα. Τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Πόσοι άνθρωποι παθαίνουν, πώς το λένε αυτό, αλσχάιμερ αυτό είναι λοιπόν που πρέπει πράγματι να το αντιμετωπίσετε και όχι τα θέματα των εμβολίων. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Τόμας Λόντγκρεν για τη θαυμάσια εργασία που έχει, εργασία που έχει κάνει σαν πρόεδρος της ΕΜΕΑ, σαν διευθυντής της ΕΜΕΑ. Σα ευχαριστώ κύριε Λέγκρεν, εξ ονόματο και όλων των συναδέλφων, για τι εξηγήσει μα σήμερα το απόγευμα. Ευχαριστώ όλου. Ε, λίγη λοιπόν η συνεδρίαση αυτή.